Uh, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε τώρα γιατί έχω και κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Αν τω μεταξύ θα έρθουν και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο τη Δευτέρα να φτάσουν όλοι στην ώρα τους, μια που ταξιδεύουμε κιόλα. Για το, το πρώτο θέμα, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Υπάρχει αντίρρηση. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία. Συνεπώ, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι η συνεδρία σε αυτή βγαίνει μέσω διαδικτύου στον ε, κυβερνοχώρο. Συνεπώς φροντίστε να πατάτε το μικρόφωνο. Κάθε φορά που πατάτε το μικρόφωνο ε, τότε η κάμερα στρέφεται σε εσά και φαίνεστε εσείς στην κάμερα. Όταν κλείνετε το μικρόφωνο τότε φεύγει από εσά η κάμερα. Βέβαια πρέπει να κάθεστε για να μπορεί η κάμερα να πιάνει το πρόσωπό σας. Αν στέκεστε όρθιοι, τότε δεν θα φαίνεται το πρόσωπό σας στην κάμερα. Δεύτερον, η ψηφοφορία που έχουμε για την ε, οδηγία μέχρι τις 27 Απριλίου αναβάλλεται η ψηφοφορία αυτή για τις απαιτήσει διαφάνειας. Αυτό για να έχουμε περισσότερο καιρό για να πετύχουμε συμβιβαστικές λύσεις η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που συμμετέχει σε αυτή την ιστορία βάσει του άρθρου 50 μπορεί επίσης να αναβάλει την ψηφοφορία της. Δεν έχουν ακόμα αποφασίσει όμως. Επίσης πρέπει να σας πω ότι θα υπάρξει ακρόαση στις 14 Απριλίου το απόγευμα για την κατάσταση στην Ελλάδα. Τις λεπτομέρειες για την ακρόαση αυτή θα τις πάρετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης, θα έχουμε και μια έκτακτη συνάντηση στις 19 Απριλίου στο Στρασβούργο, όπου ο κύριος Παπαδήμος, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα έρθει και θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση για το 2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης υπάρχουν δύο προφορικές ερωτήσεις και σχέδια ψηφίσματος για να εγκριθούν τον Απρίλιο από την Επιτροπή μας. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τις εξαιρέσεις για τα οχήματα και το δεύτερο είναι για τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική για, για το ευρώ επίσης στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Τις λεπτομέρειες θα τις μάθετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τέλος, η γραμματεία επεξεργάζεται τις 1600 περίπου τροπολογίες που έχουμε για, τις, ε, για την έκθεση για το εποπτικό πακέτο. Ελπίζω, δουλεύει η γραμματεία είπαμε έτσι, προσπαθεί να προχωρήσει. Ίσως όμως να μην μπορέσουν ε, οι ευρωβουλευτές να έχουν όλες τις τροπολογίες στις 23 του μηνός, αύριο. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι καλώς θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και άλλη φορά και τότε θα υπάρχουν οι μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες, φαντάζομαι. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που έχω να σας κάνω. Σημείο 3 τώρα στην ημερήσια διάταξη. Εδώ με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη συνεδρίασή μας τον κύριο Γιούγκερ. Γνωρίζετε βέβαια ότι είναι πρόεδρος της Ευρωομάδας και ότι έχει μια δύσκολη δουλειά. Ο κύριος Γιούνκερ θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα απαντήσει σε ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών βάσει της διαδικασίας Catch the Eye, όποιον βλέπει ο Πρόεδρος. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω εδώ ότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι στην ημερήσια διάταξη, περιμένουμε ότι κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων θα προκύψει το θέμα και ο κύριος ε, Γιούνκερ έτσι κι αλλιώς θα μας βοηθήσει για να μας εξηγήσει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς ε, θα ερχότανε, οπότε δεν θελήσαμε να το βάλουμε σαν ξεχωριστό θέμα. Εννοείται ότι θα συμπεριληφθεί. Λοιπόν, κύριε Γιούγκερ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη μου ευχαρίστηση. Σας ξαναβρίσκω σήμερα στη συνεδρία της Επιτροπής σας είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ, μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, που γνωρίζετε ότι επέφερε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία μας. και στις διαδικασίες που εφαρμόζονται στη λειτουργία της Ευρωμάδας. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας επέτρεψε στην Ευρωμάδα να αναβαθμιστεί από το άτυπο καθεστώς δηλαδή που είχε η συνθήκη το, την αναγνωρίζει και δίνει μια κάποια επισημότητα στις εργασίες του. Το πρωτόκολλο 14 παράρτημα της ε, συνθήκης ε, της Λισαβόνας προβλέπει ο πρόεδρος του, της Ευρωμάδας να εκλέγεται για δυόμιση χρόνια. Και επανεξελέγει λοιπόν από την Ευρωμάδα στις 18 Ιανουαρίου. Εγώ είχα υποβάλει πριν επανεκλεγώ, είχα καταθέσει μερικές προτάσεις ε, στους συναδέλφους που ως ε, στοιχεία, προγραμματικά στοιχεία, γύρω από τα οποία ε, έχω και ορισμένες ιδέες, τις οποίες θα σας παρουσιάσω σύντομα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωμάδα να προχωρήσει με νέο πνεύμα στις εργασίες της, ε, του συντονισμού των ε, δημοσιονομικών μας πολιτικών. Η Ευρωμάδα Η Ευρωομάδα χρειάζεται μία μεγαλύτερη δυνατότητα επαφής για τους προϋπολογισμούς. Οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να παρουσιάζουν πρώτα στα εθνικά τους κοινοβούλια και μετά να έρχονται και σε εμά να τα παρουσιάζουν και ελπίζουμε να λαμβάνουν και υπόψη όταν θα παρουσιάζουν τους προπολογισμού στην Ευρωζώνη τις παρατηρήσεις που οι συνάδελφοι από τις άλλες χώρες θα του κάνουν. Επίσης η Ευρωμάδα θα δημοσιεύει περιοδικά σημεία αναφοράς τα οποία αναλαμβάνονται υπόψη και από τους παρατηρητές και από όσους συμβουλεύονται την Ευρωμάδα για να έχουν υπόψη τους γενικότερα τις τάσει της Ευρωμάδας. Η Ευρωμάδα τις επόμενες εβδομάδες θα εξετάσει τη στρατηγική εξόδου, αυτό που ονομάζεται στρατηγική εξόδου. Εμείς έχουμε απλώς ε, βάλει μερικούς στόχους. Θα πρέπει τώρα να δούμε ποιο θα είναι το φορολογικό κίνητρο, το φορολογικό στίμουλους για να μπορέσουμε να βρούμε έγκαιρα, ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά, τη στιγμή σταθεροποίησης των δημοσιονομικών μας. Εμείς θεωρούμε ότι το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ε, την υποστήριξη των κρατών και θα πρέπει να τελειώνουμε με τα πλεονεκτήματα των τραπεζών που δέχονται τη δημόσια βοήθεια χωρίς να την έχουν ανάγκη. Θα πρέπει <coughs> να ενισχύσουμε την αγορά εργασίας και την αγορά των προϊόντων τα μέτρα τα οποία αποφασίσαμε επέτρεψαν να απαλύνουμε την ε, κρίση στην αγορά εργασίας. Αλλά αυτοί οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους ή θα τη χάσουν στο μέλλον δεν βλέπουν τα καλά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε να υποστηρίζουμε πιο έντονα την πολιτική απασχόλησης ε, είτε ε, μέσα από τη μερική ανεργία ή άλλα πράγματα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ποια θα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να σταματήσουμε βαθμία αυτά τα μέτρα υποστήριξης. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από τις ε, εθνικές ιδιομορφίες της κάθε χώρας. Εμείς λοιπόν εμπλουτίσαμε και το Σύμφωνο Σταθερότητας με μια νέα έννοια, σχεδόν νέα, που λέει ότι μέσω πρόθεσμα οι χώρες της ζώνης θα πρέπει να έχουν ένα έλλειμμα μικρότερο του 3% αλλά θα πρέπει να εξισορροπήσουν τον προϋπολογισμό τους. Βέβαια δεν ήρθε η ώρα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά αυτή η ιδέα δεν έχει εγκαταλειφθεί. Θα επανέρχεται σταθερά και συμβατά με τις πολιτικές που θα πρέπει να αναπτύξουν τα κράτη-μέλη για να εξηγιάνουν τα δημοσιονομικά τους. Βέβαια, το θέμα αυτό δεν μου φαίνεται άμεσης επικαιρότητα, οπότε δεν θα σταθώ παραπάνω Όταν εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε το ενιαίο νόμισμα πιο συλλογικά και πιο αλληλέγγυα, θα πρέπει να επεκτείνουμε το εφαρμοστικό μας πεδίο των οικονομικών πολιτικών. Οι Υπουργοί Οικονομικών έδωσαν την εντύπωση, δεν ήταν η σωστή εντύπωση, αλλά την έδωσαν, ότι, ότι ασχολούνται μόνο με τον προϋπολογισμό. Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θέτουν απαιτήσει που ξεπερνούν τις απλές δημοσιονομικές πλευρές. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, όπως κάναμε και σήμερα, στις διαφορές που διαπιστώνουμε στη νομισματική ζώνη και θα πρέπει να προσέξουμε επίσης ιδιαίτερα τις μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες έχουν ενταθεί μετά από τη δημιουργία του ευρώ και που δεν έχουν εξαφανιστεί. Εντάξει, άλλες εντυνόμενες, άλλες μειονόμενες, αλλά εκεί είναι. Οι γενικές λοιπόν ανισορροπίες ε, στην εσωτερική μας ε, ζώνη δημιουργούν όλο ένα και περισσότερα προβλήματα. Οπότε εμείς πρέπει να βρούμε τη μέθοδο για να συζητήσουμε μεταξύ μας το πώς θα γκρεμίσουμε τους φραγμούς προς την ανάπτυξη. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να συζητήσουμε για το τι μέσα θα αναπτύξουμε στην Ευρωζώνη, ούτως ώστε να αυξήσουμε την ανάπτυξη κατά την έξοδό μας από την κρίση. και επίσης να αυξήσουμε έλεγα την ανάπτυξη σε 1,5-2% τουλάχιστον, διότι άμα δεν έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, τα συνταξιοδοτικά μας ταμεία κινδυνεύουν, δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το βιωτικό επίπεδο και το κοινωνικό στάνταρ της Ένωσης. κάτι το νέο που θέλουμε, μετά από κάθε νέα συνεδρίαση της Ευρωζώνης να εξετάζουμε την θέση ε, ανταγωνισμού ενός, του ενός ή του άλλου κράτους μέλους. Εμείς ε, μέχρι τώρα δεν προσέξαμε την απώλεια ανταγωνιστικότητας της μίας ή της άλλης χώρας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μετά από κάθε συνεδρίαση θα εξετάζουμε αναλυτικά την κατάσταση μιας χώρας μέλη, μέλος. Θα ξεκινήσουμε με τις χώρες που θα είναι εθελόντρες και μετά θα περάσουμε από το κόσκινο την κατάσταση όλων των άλλων κρατών. Εμείς λοιπόν ενθαρρύνουμε ως Ευρωμάδα την Κομισιόν ε, να προσφεύγει στο άρθρο 121 της Συνθήκης που επιτρέπει την Κομισιόν να απευθύνει προειδοποίηση στο κράτος μέλος εκείνο το οποίο απομακρύνεται από τις ε, θεμελιώδεις αρχές ε, της κοινά συμφωνημένης στην Ευρωμάδα Οικονομικής Πολιτικής. Εμείς το κάναμε αυτό μία πρώτη φορά όταν εξετάσαμε την ελληνική κρίση. Ενθαρρύνουμε δε την Κομισιόν στα πλαίσια του άρθρου 136 της Συνθήκης να παρουσιάσει μία πρόταση που θα προτείνει μέσα για να εμβαθύνουμε στον συντονισμό και την παρακολούθηση των οικονομικών πολιτικών. Η νέα συνθήκη δίνει αυτές τις δυνατότητες στην Κομισιόν. Θα θέλαμε λοιπόν η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν πιο σοφά και φρόνημα αυτό το εργαλείο. Λοιπόν, για τις διαδικασίες τώρα. Εμείς δεν θέλουμε να μπλέκουμε τις διαδικασίες μεταξύ τους. Δηλαδή, τα μέσα που έχουμε και τις διαδικασίες στα πλαίσια της Ατζέντα 2020 ε, και τις ε, διαδικασίες και τα μέτρα που έχουν να κάνουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν πρέπει λοιπόν να τα μπλέκουμε όλα αυτά. Και ούτε επίσης να τα μπλέκουμε με τις άλλες διαδικασίες τις οποίες θα αποφασίσουμε να αναλάβουμε. Πρέπει λοιπόν να ορθολογικοποιηθεί η όλη λειτουργία και να δοθεί και μία ορατότητα στην Ευρωμάδα και στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε την οικονομική μας ζώνη. Δεν θεωρούμε, επειδή οι συνθήκες δεν το προβλέπουν ε, ούτε έτσι, ότι η ευρωμάδα θα ήταν ένα περιορισμένο γκρουπ ένα περιορισμένο κλαμπ. Όσοι έχουν αποφασίσει το opting out μπορούν κάλλιστα να μπουν στην Ευρωζώνη όταν θα έχουν συμπληρώσει όλα τα κριτήρια σύγκλησης και μπορούν να γίνουν μέλη. Τώρα για τις νέες προσχωρήσεις εμείς αποφασίσαμε να εξετάζουμε από καιρού εις καιρών την κατάσταση σύγκλησης των υποψηφίων χωρών για την Ευρωζώνη. Και θα το κάνουμε ε, όταν ε, η Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν θα έχουν ορίσει τα κριτήρια σύγκρισης και θα καλούμε στην Ευρωζώνη και τη χώρα που πληρεί αυτά τα κριτήρια να το συζητήσουμε μαζί της, όπως επίσης και τις υποψήφιες χώρες ε, και θα εξετάζουμε και την αηφορία με την οποία οι χώρες αυτές μπορούν να συνεχίσουν. Προς στιγμή λοιπόν τώρα, κυρία Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε... το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. και θα είμαι ιδιαίτερα ακριβής θυμίζοντας ε, στον εαυτό μου ότι θα ήταν πιο σοφό να ήμουν πιο συγκεκριμένος συγκρατημένος, συγγνώμη. Η κατάσταση της Ελλάδας είναι φανερή στους ειδήμονες που είστε εσείς. Η κατάσταση της Ελλάδας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια συνεχή απώλεια παραγωγικότητας της Ελλάδας από τη στιγμή που έγινε μέλος της Ευρωζώνης. Προς στιγμή το πρόβλημα είναι δημοσιονομικό, είναι πρόβλημα προϋπολογισμού και για να το αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις διατάξεις του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας, έτσι όπως αποφασίστηκε το Μάρτιο του 2005 και αυτό ερμηνεύεται ως εξής. Η Ευρωομάδα τον Φεβρουάριο και άλλες φορές βέβαια κάλεσαν την Ελλάδα να αναλάβει συμπληρωματικά μέτρα διότι θεωρούσαμε ότι τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης δεν ανταποκρινόντουσαν στους στόχους που έπρεπε να προσεγγιστούν. Πρέπει να σας πω εδώ ότι εντυπωσιάστηκα από το θάρρος και από τα μέτρα τα οποία ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια πολιτική που είναι αξιόπιστη και αν οι καιροί στις αγορές ήταν κανονικοί καιροί, νορμάλ καιροί, θα διασφάλιζαν λοιπόν τις, αυτές τις αγορές, αυτά τα μέτρα. Εμείς ζητήσαμε από την Ελλάδα να πάει το έλλειμμά στο 8,7% για να πληρώσει αυτό το έλλειμμα και τα μέτρα τα οποία έχει ψηφίσει η ελληνική κυβέρνηση θα επιτρέψουν να, την εξυγίανση των ελληνικών δημοσιονομικών στο χρόνο που τους αναθέσαμε, προσεγγίζοντας όλους τους στόχους που από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση ορίσαμε. Διαπιστώνω λοιπόν ότι η Ελλάδα πήρε πολύ καλά μέτρα σε μια πρώτη φάση, σε το αίτημα που υποβάλαμε, στο δεύτερο αίτημα πήρε και άλλα μέτρα. Πήρε τα μέτρα που έπρεπε, το Κοινοβούλιο της Ελλάδας ενέκρινε αυτά τα μέτρα. Η Ελλάδα λοιπόν σέβεται απόλυτα το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Επιπλέον, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να το επιβάλλουμε να ακολουθήσει αυτόν το δρόμο των μεταρρυθμίσεων, πράγμα το οποίο έκανε ο ικανότατος άνθρωπος ο οποίος προεδρεύει της ελληνικής κυβέρνησης και άμα δεν είχε ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες θα έπρεπε κάθε φορά που λαμβάνει τα μέτρα να έρχεται να απολογείται στην Ευρωζώνη. Αληθεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωζώνη υποχρεώνουν τον Έλληνα πολίτη σε προσαρμογές ιδιαίτερα επίπονες. Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό θα επιτρέψει στην Ελλάδα να βρει την δημοσιονομική της υγεία, να βρει το δρόμο της ανάπτυξης και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας η οποία δεν είναι καθόλου σε φόρμα. Εγώ Στις ε, ερωτήσεις ε, που θα μου απευθυνθούν θα κοιτάξω να απαντήσω λεπτομερέστερα. Και δεν θα μπω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά με μία λέξη. Αν η Ελλάδα χρειαστεί την βοήθεια της Ευρωζώνης, δεν θα την εγκαταλείψουμε. Η Ελλάδα εγκρίνοντας τα μέτρα τα οποία ενέκρινε, υπέδειξε την έντονη ευρωπαϊκή της βούληση να παραμείνει αξιόπιστος εταίρος της Ευρωζώνης. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να εγκαταλείψουμε στη μέση του δρόμου την Ελλάδα. Αν οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν αντιδράσουν κατά το ευκταίο στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού και συνεχίσει όλη αυτή η διαδικασία ε, κέρδοσκοπίας τότε η Ευρωζώνη θα πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη ενδιαφερόμενη χώρα. Αν εμείς κάνουμε μεγάλα λάθη χειρισμού, αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλες δύσκολες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν όταν είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Ελπίζω να μην έρθει αυτή η στιγμή. Διότι το πρόγραμμα εξυγίανσης των οικονομικών της Ελλάδας μου φαίνεται πάρα πολύ αξιόπιστο και θα προσεγγίσει τους στόχους που έθεσε σε αυτήν η Ελλάδα. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε ένα μέσο στα χέρια μας για τη βοήθεια προς την Ελλάδα για να διασφαλίσουμε και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Θυμάστε τι υπόθηκε στις, στο Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου όπου αναφέραμε την πεποίθησή μας να βοηθήσουμε την Ελλάδα αν χρειαστεί. Η Ελλάδα δεν ζήτησε βοήθεια. Το πρόγραμμα της χώρας είναι αξιόπιστο αν όμως η κατάσταση χειροτερεύσει ή αν η Ελλάδα χρειαστεί την βοήθεια όλων μας, εννοείται ότι θα οργανωθεί αυτή η βοήθεια όταν και όπως χρειάζεται. Εμείς στα πλαίσια της Ευρωμάδας προχωρήσαμε σε μια αναλυτική τεχνική συζήτηση για το μέσο το οποίο θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας αν ποτέ χρειαστεί. Δεν λάβαμε επίσημη απόφαση, διότι αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εμείς στην ε, Ευρωμάδα εκτελούμε τις εντολές που μας δίνονται από το Συμβούλιο. Και από τις 11 Φεβρουαρίου και μετά συνεχίζουμε να εξετάζουμε ένα σωρό τεχνικό ζητήματα. Και όταν θα χρειαστεί, αν ποτέ χρειαστεί αυτό το μέσο, θα το έχουμε. Δεν θα μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες για να σας ε, ανακοινώσω ποιο θα είναι αυτό το μέσο που θα θέλαμε να είχαμε στη διάθεσή μας. Το Συμβούλιο αυτήν τη εβδομάδα θα πρέπει να αποφασίσει αλλά εμείς από τεχνικής πλευράς πρέπει να τα έχουμε όλα ρυθμισμένα αν ποτέ χρειαστεί αυτό το μέσο. Εγώ αποκλείω την απριόρι συμπαθητική ιδέα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μέσο στη διάθεσή μας που όπου μάλλον θα εγγιόντουσαν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τα δάνεια που θα θυνόντουσαν στην Ελλάδα. Είναι δύο χώρες εξάλλου που το απέκλεισαν 100% αυτό το μέσο. Οπότε δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω τις εργασίες μου προς μια κατεύθυνση που ξέρω ότι δεν θα ε, οριμάσει ποτέ. Και ξέρω ότι γύρω από αυτό δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ συμβιβασμός. Οπότε θα ήταν καλό το μέσο αυτό να οργανώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη διμερή βοήθεια που θα μπορούσε να δοθεί στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να πούμε εδώ ποια θα είναι όλα, και θα είναι όλες οι λεπτομέρειες αυτού του μέσου που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ε, απασχολεί πολλές ε, καγκελαρίες. Εγώ δεν είμαι υπέρ προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορούμε να προσφύγουμε σε δύο τύπων μέσα. Διημερή βοήθεια προς στην Ελλάδα και προς. Η άλλη είναι προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια όλα τα τεχνικά τύπια ακόμη δεν τα ξέρουμε, αλλά μπορούμε κάλλιστα να προσφύγουμε σε αυτήν την διπλή ενίσχυση. Δηλαδή ένα τμήμα της βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ένα άλλο τμήμα από την ομάδα της Ευρωζώνης. Είναι όμως ακόμα πολύ νωρίς να κλείσει αυτή η συζήτηση. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε γρήγορα. Τώρα εμένα η δική μου προσωπική θέση είναι να πω ότι η Ευρωζώνη θα έπρεπε να είναι ικανή από μόνη της να λύνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη δική της ε, σφαίρα. Βέβαια δεν θα αρχίσω να, να φωνάζω σκάνδαλο σκάνδαλο άμα γίνει προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά κυρία Πρόεδρε, γρήγορα, μερικά από τα πράγματα που ήθελα να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Right, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάνω από 12 συναδέλφους που έχουν στήσει το λόγο και βλέπω ότι και άλλοι ενδιαφέρονται. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να είστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι. Θα περιοριστούμε παρακαλώ στο ένα λεπτό, θα χρησιμοποιήσω και το ρολόι. Πρώτα ακούμε τον Ζαν Πολ Γκοζέ συντονιστή για το ΕΛΚ. Παρακαλώ, Ζαν Πολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα λόγια σας. Σας παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον. Αν μου επιτρέψετε, δεν θα διατυπώσω ερώτηση, αλλά παρατήρηση. Με καλύπτουν αυτά που λέτε, αλλά πρέπει να επισημάνω επίσης ότι ο Ευρωπαίος, ο συμπολίτης μας, δεν καταλαβαίνει πια τίποτα. Οι εφημερίδες μεταφέρουν τη μία φράση των δηλώσεων από εδώ και την άλλη από εκεί. Όταν μιλούν ε, οι υπουργοί στο Συμβούλιο των Υπουργών κάνουν δηλώσεις πολύ επιφυλακτικές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όταν πρέπει για λόγους προεκλογικούς της Βρετανίας Φερρυπίν, εάν χρειαστεί, καθυστερεί η οδηγία Διεθνής Νομισματικό Ταμείο και τότε στις εφημερίδες εμφανίζεται με επιχαίους τίτλους ότι η Ευρώπη παρακολεί την εξέλιξη των δημοσιονομικών αγορών κτλ. Και εσείς μιλήσατε κιόλας για την άμυνα απέναντι στις ε, κερδοσκοπικές πιέσεις. Εγώ λοιπόν ερωτώ, και εγώ προέρχομαι από μια περιοχή της υπαίθρου, απλή ζωή, ήρεμοι άνθρωποι. Προσπαθώ λοιπόν να του εξηγήσω, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ, πως είναι δυνατόν να κάνουμε μεγάλες δηλώσεις μεγαλοσχήμονες ε, δηλώσεις για λύσεις μέσα στα δύο-τρία χρόνια. Και ερωτώ, κύριε Πρόεδρε, το εξή. Τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε τα μηνύματα που θέλετε να αποστέλλετε να γίνονται κατανοητά, ευχερέστερα και όλοι αυτοί από τις διάφορες χώρες οι οποίες διοχετεύουν καθημερινά στον τύπο πληροφορίες οι οποίες προκαλούν μόνο σύγχυση και αναστάτωση, πώς, πώς νομίζετε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Γιατί τελικά η Ευρώπη ίσως βρίσκεται σε χειρότερη θέση τώρα από ότι ήταν μέσα στο χειρότερο σημείο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Απάντηση. Συμφωνώ αρκετά μαζί σας. ότι ήδη δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυσκολία, ο πολίτης δεν μπορεί να μας παρακολουθήσει για το ζήτημα της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών και των ε, hedge funds δεν θα μιλήσω, επιτρέψτε μου, είναι ζήτημα του ΕΚΟΦΗΝ, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ. Απλώς, όπως είπατε και εσείς, διαπιστώνω με λύπη μου ότι δεν μπόρεσε το ΕΚΟΦΗΝ στις 16 Μαρτίου να προσδιορίσει μια σαφή, μια απερίφραστη τοποθέτηση ως προς τα hedge funds. Όπως θα θέλαμε ασφαλώς όλοι να δούμε. Υπήρχε μια ελπίδα ότι θα υπάρχει περισσότερη πρόοδος προς την αυτορύθμιση των αγορών, ούτε αυτό όμως μπόρεσε να προχωρήσει. Η Ισπανική κυβέρνηση ήλπιζε ότι θα μπορούσε να το προωθήσει. Δεν εξασφαλίστηκε αυτή η πρόοδο, Αλλά ασφαλώ εάν ένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη δεν μπορεί να ακολουθήσει τι συνενετικέ λύσει. δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή η ομοφωνία, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και βέβαια με δυσφορία μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε να ετοιμαστούν οι πάντε να ακολουθήσουν του ρυθμού τη Ευρώπη της, της πλειοψηφίας. Για την ε, Eurogroup και την Ελλάδα. Το μήνυμα είναι σαφές νομίζω. Η Ελλάς υιοθέτησε ένα φιλόδοξο και αξιόπιστο πρόγραμμα ένα πρόγραμμα το οποίο οφείλει, πρέπει να πείσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εάν αυτές δεν πιστούν, επειδή έχει ξεκινήσει μεγάλη κερδοσκοπική ε, επίθεση αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, θα πρέπει και η Ελλάδα να είναι σε θέση να προχωρήσει με ένα μέσο το οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε σήμερα και να αποφασίσουμε ενδεχομένω, αλλά την ώρα που θα χρειαστεί θα αποφασιστεί. Η Ελλάδα ασφαλώ θα πρέπει να προχωρήσει σε κάθε προσπάθεια που της ανήκει, που είναι δικών της καθήκον, θα πρέπει να κάνει δηλαδή το δικό της καθήκον για να προχωρήσει, να βγει από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα αυτονόητο είναι και το καθήκον της αλληλεγγύης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι βλέπουν οι πολίτες της Ευρώπης ξεκάθαρα την εικόνα. Η Ελλάδα κάνει ό,τι έχει να κάνει και δεν την εγκαταλείπουν οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν εσείς στη δική σας την εκλογική περιφέρεια έχετε μια διαφορετική εικόνα, εκεί που ε, ξέρω εγώ τουλάχιστον ότι ο κόσμος έχει κοινή λογική, απλή κοινή λογική και ίσως ε, να μην ε, αμφισβητεί την καλή λογική και των δικών μας των επιλογών. Νομίζω ότι θα αναγνωρίσει ότι ήταν σωστές οι επιλογές μας και φρόνιμες. Ο κύριος Ούντε Μπούλμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, τρεις τι ερωτήσει πολύ σύντομε, πώ να τι τετυπώσω πιστεύω, σύντομα σε ένα λεπτό. Μιλήσατε για ένα μηχανισμό που διαμορφώνεται, μα έχει όμω μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 153, το οποίο δεν εφαρμόζεται εδώ γιατί ε, αφορά τα, τα κράτη εκτό τη Ευρωζώνη. Υπάρχει όμω ε, η δυνατότητα τη οικονομική παρέμβαση εδώ που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει ε, ή μάλλον να διαθέσει πιστώσεις λογικές στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω εάν εδώ θα υπαχθούμε στο 152, στο 136. Δεν καταλαβαίνω όμω γιατί σιωπά αυτό ο οργανισμό. Είναι ένα οργανισμό ο οποίο μέχρι τώρα θεωρούσα, τουλάχιστον εγώ, ότι ήταν αρκετά ε, λογικό και οικονομικό στη χρήση του και για τα κράτη-μέλη. Γιατί λοιπόν να μην προχωρήσει σε εφαρμογή. Επίση υπάρχουν κάποιοι που μιλούν για έξοδο από την Ευρωζώνη. Είχα την εντύπωση, εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα, ότι τα νέα κράτη-μέλη ήταν λίγο πολύ υποχρεωμένα να ενταχθούν στο ευρώ και ότι ήταν λίγο πολύ μέρο του ευρωπαϊκού κεκτημένου το ευρώ. Είναι λοιπόν δυνατόν νομικά να λέει κανείς ότι μπορεί, μπορεί να αποχωρήσει από, ένα, ε, από την Ευρωζώνη ένα κράτος μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από το ευρώ. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ε, να ενταθεί περισσότερο η εκ των προτέρων επιτήρηση, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις δεσμενέστερες επιπτώσεις των, ε, της εκ των υστέρων μόνο αντιμετώπιση των προβλημάτων ο κύριος Γιούνκερ. Κύριε συνάδελφε, κύριε Μπούλμον. Το μέσον το οποίο από ό,τι φαίνεται θέλετε εσείς να εφαρμοστεί είναι προφανές ότι δεν την χάνει της υποστήριξης όλων των κρατών μελών. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό σύντομα. Θα πρέπει να βρούμε όμως ένα μέσον τώρα εμείς, δηλαδή δεν έχουμε περιθώριο να καθυστερήσουμε περισσότερο αναζητώντας συνενέσεις εκεί όπου δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναστήσουμε ενδεχομένω άλλα μέσα. Και επίση θα πρέπει να σα πω ότι για μένα το 122 νομική βάση δεν, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δηλαδή ούτε φυσική καταστροφή έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ούτε άλλα προβλήματα, άλλου τύπου προβλήματα. Έχουμε να κάνουμε ένα κράτος το οποίο είναι χρεωμένο. Αυτό είναι το πρόβλημα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την εφαρμογή του άρθρου 122 και να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά μέσα για την ε, αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή για διμερή θελοντική ε, βοήθεια όπως έχουμε με τα τρίτα κράτη της Ευρώπης. Ε, τα τρίτα κράτη έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κράτο μέλο, έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία έχει λάβει σωστέ αποφάσει και θα είναι πιστική πιστεύω ε, ω προς τις επιλογές της και ως προς το πακέτο μέτρων που εισάγει για να εξηγιάνει τον προπολογισμό της. Υπάρχει από τον κύριο Σόιμπλε, τον Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας, ένα ερώτημα το οποίο ετέθη για συζήτηση, αν υπάρχει ανάγκη για ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Το ερώτημα αυτό πρέπει να σας πω ότι με έχει απασχολήσει πολύ. Το έχω συζητήσει, το έχω μελετήσει. Η περίπτωση της Ελλάδας μας δείχνει ότι δεν έχουμε ικανό μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανό εργαλείο αν θέλετε, το οποίο να μας επιτρέπει ε, αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουμε ε, μια τέτοια οικονομική κρίση. Αλλά ούτε και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα ήταν μια ικανή λύση πιστεύω, γιατί η κρίση στην Ελλάδα είναι μια βαθιά κρίση, είναι μια κρίση που χρειάζεται άμεση απάντηση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μέσο το οποίο μόνο μέσο πρόθεσμα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί. Γι' αυτό και λέγω ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητήσουμε την εισαγωγή ενός μεσοπρόθεσμου μέσου. Μπορώ να το συζητήσω, είναι ένα θέμα το οποίο μπορώ να κάτσω και να συζητήσω στις τράπεζες των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν με έχει πείσει η προοπτική αυτή. Και γιατί δεν με έχει πείσει, διότι επίσης πιστεύω ότι αν προβλεφθεί η δυνατότητα του αποκλεισμού ενός κράτους, θα πρέπει ταυτόχρονα να προβλεφθεί και η δυνατότητα της αποχώρησης ενός κράτους. Άρα, της εκούσης αποχώρησης δηλαδή. Άρα, ίσως θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες και πώς μπορούμε να διακρίνουμε την εθελοντική αποχώρηση ή τον αποκλεισμό ενός κράτους. Πράγμα το οποίο θα μας φέρει οριστικά και αμετάκλητα σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε γιατί θα είμαστε πια όχι εμεί εκείνοι οι οποίοι θα ορίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά εκείνοι οι οποίοι θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις αμέτωχοι κατά πάσα πιθανότητα και θα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν θα έχουμε δηλαδή την δυνατότητα να κινηθούμε για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα την ώρα που εμφανίζονται. Νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και για την Ένωση και για το κράτος βέβαια το ίδιο το οποίο ενδεχομένω αποκλειστεί και το οποίο δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του καθόλου εύκολα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο σκόπιμο να εντείνουμε την, ε, τις διατάξεις και το σύστημα της εκ των προτέρων παρακολούθησης και επιτήρησης ενός κράτους έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, έτσι ώστε να προλάβουμε δυσμενείς εξελίξεις που θα μας φέρουν ενώπιον ε, ή μέσα καλύτερα σε μια κρίση. Ευχαριστώ κυρία Γκρινλάρτ. Όπως και ο κύριος Ογκοζές, συμφωνώ με την παρατήρηση που έκανε. Επιτόπου τελικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια τίποτα. Και όταν ακούμε και χάρηκα που σας άκουσα να το λέτε ότι δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα στην τύχη της. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε. Αλλά όταν συγχρόνως ακούμε διαδόσεις που μιλάνε ότι μπορεί να βγει μια χώρα μέλος, καταλαβαίνετε ότι ο Ευρωπαίος πολίτης τα χάνει. Εσείς λοιπόν που συνεισφέρετε στη δημιουργία του ευρώ, τι μήνυμα μπορείτε να δώσετε σε αυτούς που κοιτάνε τις διάφορες στατιστικές, ε, τα διάφορα στοιχεία και που ίσως τότε δεν θα καταλήγαμε σε ενιαίο νόμισμα, αν το είχαμε κάνει τότε. Τώρα λοιπόν υπάρχει θέμα εσωτερικής αξιοπιστίας. Τότε δεν θα έπρεπε να αναλάβουμε εξωτερικά μια πρωτοβουλία. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτή την ιδέα για να δείξουμε και στον πολίτη ότι υπάρχει βούληση να συνεχίσουμε μαζί και ότι η βούληση αυτή είναι πιο ισχυρή από τις δυσκολίες. Κατά τα άλλα, για την Ελλάδα σας έχουμε εμπιστοσύνη. Ετοιμάστε όμως καλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Μπορούμε να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να είναι χρήσιμο. Να υπάρχει και μόνο. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα να σας απαντήσω τελικά, λέει ο κύριος Γιούνκερ. Γαλλικά ή γερμανικά. Μια που χρησιμοποίησατε και μια γερμανική έκφραση. Δεν ξέρω ποιος θα καταλάβει τελικά. Αν σα μιλήσω Λουξεμβουργέ και θα μα καταλάβει κανεί άλλο. Ναι, όχι, εγώ εξασκούμε με την κυρία Λούλινγκ όμω. Μην ανησυχείτε, λέει κυρία Κουλάχ. Καλώ. Α μιλήσω λοιπόν γερμανικά. Νομίζω ότι μόνο οι Λουξεμβούργοι θα είναι σε θέση να μα καταλάβουν, γι' αυτό ίσω είναι καλύτερα να βρω μια άλλη γλώσσα, να επιλέξω μια άλλη γλώσσα. Δεν ε, μπορώ παρά να πω ότι έχουν δίκιο όσοι κάνουν τη διαπίστωση ότι οι παρατηρητέ και αυτοί οι οποίοι μας εκπροσωπούν, δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τη συζήτηση όλη αυτή που γίνεται γύρω από την Ελλάδα. Εγώ θέλησα να συνεισφέρω στη σαφήνεια και γι' αυτό και είπα ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει όλες τις προσπάθειες που χρειάζεται και ότι είναι αξιόπιστες οι προσπάθειες αυτές και αρκετές και αν αποδειχτεί ότι δεν αρκούν, τότε η Ευρωζώνη πρέπει να απαντήσει με αλληλεγγύη και ότι δεν χρειάζεται μέσα στα πέντε λεφτά να αποφασίσουμε τι και πώς. Η Ελλάδα δεν ζήτησε στήριξη, η Ελλάδα δεν κινδυνεύει με πτώχευση αυτή τη στιγμή, οπότε δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε για τις λεπτομέρειες του μέσου που θα χρησιμοποιήσουμε για να τη στηρίξουμε. Είπαμε ότι αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Τώρα η εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης. Πολύ συχνά έχω αναφερθεί στα συστατικά μιας τέτοιας ιδέας. Υπάρχουν όμως αντιστάσεις, μεγάλες αντιστάσεις, γι' αυτό και δεν προχωράμε αρκετά. Αντιστάσεις για αυτήν την ε, εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης. Η Επιτροπή, δίχως άλλο, χρησιμοποιώντας τις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας, θα φροντίσει να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για μια τέτοια εξωτερική εκπροσώπηση που να είναι πιο συνεκτική από αυτήν που έχουμε τώρα εμείς. Γιατί είναι, αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία. Λείπει ομοιομορφία. 14 ομιλητέ, λέει πρόεδρο, έχω ακόμα. Οπότε προτείνω το εξή. Σβέν Κιγκολτ, πρώτα απ' όλα, μια που είναι συντονιστή από του πράσινου. Δεν έχω άλλο συντονιστή στον κατάλογο. Οπότε μετά θα ξεκινήσω με τι ομάδε. Και ο κύριο Χουντή, ναι. Σβέν. πρότεση. Κύριε Γιούνκερ, εγώ μπορεί να μην πήγα το Σαββατοκύριακο στην ε, Γαλλία, στην Ήπεθρο της Γαλλίας, αλλά ήμουν στην Αθήνα, σε μια εκδήλωση με πολλές ομιλίες και πρέπει να σας πω ότι επιστρέφοντας ήμουν πολύ πιο ε, απεσιόδοξος από ότι πηγαίνοντας. Μιλήσατε για το πρόγραμμα εξυγίανσης ελληνικής κυβέρνησης, ότι είναι ένα καλό ε, και αξιόπιστο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες πολίτες διαφωνούν μαζί σας. Και να σας πω γιατί. Από ό,τι είδα εγώ, ο κύριος λόγος που διαφωνούν είναι ότι τα τελευταία 10-20 χρόνια εκείνοι οι οποίοι εξασφάλισαν τα μεγαλύτερα έσοδα κέρδισαν δηλαδή τις μεγαλύτερες περιοδοσίες, τις κέρδισαν παράνομα, είτε από δωροδοκία, είτε δηλαδή ε, γιατί δεν χρειάστηκε να πληρώσουν ποτέ κανένα λογαριασμό και κανένα σπασμένο και ως εκ τούτου είναι αυτοί οι οποίοι δεν ε, τηρούν ουσιαστικά και τις συνθήκες της ε, Λισαβόνας και ως εκ τούτου το πρόγραμμα της εξυγένσης της κυβέρνησης δεν αντιστοιχεί στα όσα υποτίθεται ότι θα πρέπει να τηρήσει δηλαδή τη συνθήκη τη Λισαβόνας η εξυγίανση σημαίνει ότι θα υπάρχει μια εξυγίανση του προπολογισμού, ότι θα πρέπει δηλαδή να εισαχθεί η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και ε, ότι θα διαραγούν τα κοινωνικά προνόμια ε, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται στο απειρόβλητο. Ερωτώ λοιπόν ποια είναι η θέση στην υπόθεση αυτή και στη συζήτηση και μέσα στο Eurogroup ενδεχομένω, ποια είναι το μήνυμα που αποστέλλεται, που στην ελληνική κυβέρνηση. Για εκείνου που δωροδοκήθηκαν, για εκείνου που έδωσαν ε, ρουσφε, ε, βαξίσια, τι έχετε να πείτε, πώ αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε και ο ελληνικό πληθυσμό τη Ελλάδα, ο Έλληνα πολίτη να μην έχει την οειδεύουν και τελικά μόνο αυτό καλείται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Απάντηση. Γιούνκερ. Δική μου δουλειά δεν είναι το να κρίνω εάν είναι η εσωτερική κατανομή του βάρους δίκαιη ή μη. Αλλά βέβαια μπορώ να έχω άποψη. Έχουμε καλέσει τους Έλληνες συναδέλφους και αυτό από πολλές πλευρές να κοιτάξουν το πράγμα από πολλές οπτικές γωνίες και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαρθρωτικές δηλαδή μεταρρυθμίσεις τους έχουμε καλέσει και σε φορολογική δικαιοσύνη. Έχουμε πει δηλαδή ότι η φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να επιβαρυνθούν ανάλογα με την κατάστασή του ο καθένας και με τον βαθμό στον οποίο έχουν συμβάλει σε αυτή την τόσο κακή κατάσταση από τους Έλληνες συναδέλφους με τους οποίους έχω συνομιλήσει και μιλώ για ανθρώπους διαφορετικών επιπέδων και αξιωμάτων, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια σημαντική πρόοδος ως προς την ε, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολόγησης, δηλαδή της αναλογίας του φόρου. Έχει κριθεί δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η αναλογία η φορολογική που υπήρχε. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όντως αυτό να ισχύει. Δηλαδή, όποιος έχει πιο φαρδείς ώμους να σηκώνει και μεγαλύτερο βάρος, όπως λέμε. Είναι γνωστό ότι έχει κενά το ελληνικό φορολογικό σύστημα, από τα οποία μπορεί κανείς να ξεφύγει και είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βρει τον τρόπο να καλύψει αυτό το πρόβλημα. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τέσσερις ομιλητές και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Χουντή, ο οποίος μιλάει εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. μετά Σαλαβράκος και μετά ο κύριος Γιούγκερ προηγουμένως η κυρία Ινφέλτ επίσης. αναλυτικά ελληνικά μιλάω, αναφερθήκατε αναλυτικά στην περίπτωση της Ελλάδας, ενώ γνωρίζετε ότι υψηλά ελλείμματα, υψηλό χρέος και απώλεια της ανταγωνιστικότητας από 10 ως 20% είχαμε και σε άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα όταν μπήκαν στην Ευρωζώνη. Η ερώτηση εδώ είναι, έχετε προβληματιστεί για την ορθότητα του Συμφώνου Σταθερότητας. Έχετε προβληματιστεί μήπως υπάρχουν δομικά προβλήματα στην Ευρωζώνη. Και δεύτερο, μιλάτε για μορφή αλληλεγγύης, ένα μηχανισμό βοήθειας και στήριξης της Ελλάδας. Έχετε παρακολουθήσει όποτε εσείς, ο κύριος Τρισέ, άλλοι αξιωματούχοι, κάνετε δηλώσεις αντιφατικές, οθείτε και αυξάνεται η κερδοσκοπία με συνέπεια τα θαραλέα, όπως είπατε, μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση, σκληρά κατά τη γνώμη μου, σε βάρος των εργαζομένων, να εξανομίζονται από, το από τον κογλυφικό δανεισμό. Και το τελευταίο, όσο αφορά την πιθανότητα προσφυγής της Ελλάδας ή και ενδεχομένως και άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπατε ότι είσαστε αντίθετο. Τι δουλειά λοιπόν έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ήδη έχει μπει στην αυλή της Ευρωζώνης καθώς εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν στην Επιτροπή που επιθεώρησε τα οικονομικά της Ελλάδας, εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι στην Επιτροπή που επιτηρεί την προσπάθεια κάλυψης των ελλημάτων. Astrid. Astrid. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Γιούνκερ για την παρουσίασή του. Πολύ ιδιαίτερα πλούσια ήταν. Και εγώ, όπως ε, και ο κύριος Γιούνκερ, ε, κοιτάζω με θαυμασμό αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα ε, και τα μέτρα που έχει αναλάβει. Εγώ ξέρω και να έχουν το κουράγιο να εξηγιάνουν έγκαιρα τους προϋπολογισμούς τους. Αλλά βέβαια αυτό το αφήνω στον κύριο Γιούνκερ να ασχοληθεί αυτός. Εγώ έχω μία ερώτηση σχετικά με το μέσον. Διότι είπατε δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να χαθεί, δεν θα την αφήσουμε στην τύχη σας αποκλείσατε εσείς ε, την εγγύηση των δανείων από, από τα κράτη-μέλη, γιατί είπατε είναι μερικοί που δεν θέλουν. Αλλά είπατε ότι οργανώνονται διμερείς ε, προσπάθειες ενισχύσεις. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά τώρα, άμα πούμε μια χώρα σαν τη Γερμανία δεν θέλει να συμμετέχει ως εγγυητής ε, τι θα γίνει, θα ήταν ας πούμε θα έδινε διμερή βοήθεια, θα συμμετείχε, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Ή έχετε τη γνώμη ότι δεν θα συμμετέχουν όλοι. Και ξέρετε τώρα και όλοι αυτοί, αυτό το μπρούχαχά, η κακοφωνία τέλος πάντων, όπου έχουμε διαψεύσεις, δηλώσεις, κόντρα διαψεύσεις κλπ. Ε, τώρα πια σε αυτήν την κακοφωνία η κυρία Λαγκάρντα εκουσίως ταράζει τα νερά ασκώντας κριτική στη γερμανική οικονομική πολιτική λέγοντας ότι αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Γερμανία διότι έχουν την εντύπωση ότι είναι ο κακός μαθητής που κάνει κριτική στον καλό μαθητή ότι δεν έφυγανε σωστά τα μαθήματά του. Από την άλλη μεριά όμως ένα σωρό οικονομολόγοι λένε ότι τελικά η Γερμανία είναι αυτή η οποία εκμεταλλεύεται την αγοραστική δύναμη των γειτόνων της από τη χρήση του ευρώ. Λοιπόν, η κυρία Λαγκάρντ ίσως θα μπορούσε να έχει και άδικο και δεν είναι και στην ιδανική θέση να το πει. Τι έχετε εσείς να πείτε για μια τέτοια συζήτηση η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανώδυνη διότι έχει να κάνει με το γενικότερο προσανατολισμό, το θεμελιώδη προσανατολισμό της Νομισματικής Ένωσης. Ο κύριος Καραβάκος. Ε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω ένα προβληματισμό και σε εσά αλλά και σε όλους τους συναδέλφους. Αναρωτιέμαι αν η Νέα Ορλεάνη που είναι η φτωχότερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα οικονομικό, η επιτόπου κυβέρνηση, κατά τόπου κυβέρνηση, πώς θα το έγινε. Θα αφήνεται από την κεντρική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έρμεως τους κερδοσκόπους. Πιστεύω πως όχι. Άρα πιστεύω ότι συνολικά το θέμα δεν είναι θέμα Γερμανίας ή θέμα Γαλλίας αλλά θέμα του συνόλου σαν νομικού προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσει το θέμα της Ελλάδος που στο κάτω-κάτω εγώ θεωρώ ότι είναι προσχηματικό διότι η Ελλάδα αντιστοιχεί στο 2% της οικονομίας της Ευρωζώνης. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα που πριονίζει τόσο την ενότητα όσο και τη συνοχή του ευρωπαϊκού νομίσματος. Είναι λοιπόν σαφές ότι παράλληλα με την δημιουργία ενός αδύναμου δολαρίου που έγινε στην παρελθούσα πενταετία γίνεται προσπάθεια τώρα της δημιουργίας ενός αντίστοιχου αδύναμου ευρώ. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα crash test. Ένα crash test τόσο στις αντοχές του ευρωνομίσματος αλλά κυρίως στις προθέσεις των ηγεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν αν πράγματι αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή και ένωση της Ευρώπης το έχουμε αντιληφθεί ή δεν το έχουμε αντιληφθεί. Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά, εγώ θα σας ερωτούσα ποια μέτρα προτίθεστε να εισηγηθείτε εσείς σαν Eurogroup σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή τους άλλους φορείς για τη διασφάλιση της σοβαρότητας του ευρωπαϊκού νομίσματος. Διότι αυτό για μένα είναι το θέμα, δοθέντως ότι όπως γνωρίζετε από το Σεπτέμβριο έχουν αρχίσει κουβέντες για την αντικατάσταση και του ευρώ και του δολαρίου στις διεθνείς αγορές με το ευρωκινέζικο νόμισμα, με διάφορους συνδυασμούς νομισμάτων κτλ. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι, μήπως δεν έχει γίνει αντιληπτό στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η αδυναμία του νομίσματος να αντιμετωπίσει τους κερδοσκόπους θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη εκτός αν δεν την θέλουμε νομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Sophie yes, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ για αυτά που άκουσα από τον κύριο Γιούγκερ για την αναγκαιότητα που υπάρχει να στηρίξουμε την Ελλάδα. Συμφωνώ επίσης και με τις απόψεις σας για το κατά πόσο είναι επιθυμητό ή όχι πιο πολύ παρά ε, να το πούμε σαν προτίμηση για λύση. Ναι, λοιπόν, να στηρίξουμε την Ελλάδα, αλλά όπως και κάποιοι προλαλήσαντες, δεν θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα είναι μόνο το θύμα, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει επίσης να ερευνήσει τα γεγονότα, να δει γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και αν υπάρχουν κάποια παραπτώματα που οδήγησαν σε αυτά. Πάντως συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ως προς το εξής. Το να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει να δούμε την ευρύτερη εικόνα. Γιατί στην ουσία η Ελλάδα είναι το σύμπτωμα ενός προβλήματος. Και το πρόβλημα είναι η αδυναμία του συστήματος. Το γεγονός ότι έχουμε κανόνες, έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας, χωρίς να μπορούμε ή χωρίς να έχουμε τη βούληση να το θέσουμε και σε εφαρμογή. Άρα λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός αυτό. Δεν μπορεί να λέμε ότι ναι, μια μικρή χώρα ε, αυτοί να δείχνουμε πάντα με το δάχτυλο και να λέμε ότι αυτήν τα δημοσιονομικά φταίνε. Τι θα γίνει όταν ε, κοιτάξουμε τι γίνεται με άλλες χώρες πιο μεγάλες που ξανά και ξανά ε, παραβιάζουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Το να κάνουμε πιο αυστηρό το Σύμφωνο Σταθερότητας, να είναι δηλαδή πιο δεσμευτικοί οι κανόνες και σε ακραίες περιπτώσεις να αποφασίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στον εθνικό προπολογισμό, ακόμα και εξάντε, όπως είπατε. Με ερωτηματικό το βάζω αυτό. Γίνεται. Είναι περίεργο γιατί δεχόμαστε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ελέγχους στον εθνικό προπολογισμό χωρών, αλλά όχι από εμά. Αυτό δεν είναι σε αντίφαση με την ίδια τη φύση της, ε, των κανόνων μας. Το σύστημα συντάξεων δεν μπορέσαμε να το μεταρρυθμίσουμε. Μήπως θα έπρεπε αυτό να κοιτάξουμε συγχρόνως με την περίπτωση Ελλάδα. Ο κύριος Γιούνκερ για να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοί μας δίνουν την εντύπωση ότι κάνουν μία ερώτηση. Αλλά άμα τους προσέχει κανείς από κοντά 20 ερωτήσει ο καθένας βάζουνε και πρέπει να απαντήσω σαν να ήταν τέσσερι. Ένα από τους συναδέλφου επανήλθε στο θέμα των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Δεν θέλω να πω και πάλι ότι ε, με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ εντατικά παρακολουθούμε το θέμα των στρέβλωσεων του ανταγωνισμού συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων αυτής της συγκεκριμένη υπόθεσης. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί διαρκώς στο, ε, στη ζώνη ε, ευρώ, στη Eurogroup. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις ανταγωνισμού, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα διατυπώνουμε συστάσεις και για συγκεκριμένα κράτη όταν χρειάζεται το πράξαμε άλλωστε και στην προηγούμενη μας συνεδρίαση. Απλώς δεν δημοσιεύσαμε τη σύσταση προς το συγκεκριμένο κράτος. Πήγε δηλαδή στην κυβέρνηση μόνο η εν λόγω σύσταση και όχι στον τύπο. Και από εκεί και πέρα η κάθε κυβέρνηση έχει να κάνει τη δουλειά της. Το Λουξεμβούργο κάνει ό,τι οφείλει, όπως όλες οι κυβερνήσεις πιστεύω, ένα ζήτημα πραγματικού συντονισμού των μουσουλμανικών μέσων, για το Διεθνές Ταμείο, για να ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ. Όπως έχω ήδη πει, δεν υποστηρίζω την προσφυγή στο Διεθνές Ταμείο για τη λύση του προβλήματος Ελλάδας. Πιστεύω ότι η Ευρωζώνη η ίδια είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα. Και εάν είχε πρόβλημα η πολιτεία της Καλιφόρνια, λέει ο μιλητής. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε πάλι δεν θα προσέφευγαν στις, ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απλώς θέλω να πω ότι και εμείς το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ίσως να είναι το μόνο το οποίο να θεωρεί ότι θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας. Εμείς θα πρέπει να το κοιτάξουμε και κατά αποκλειστικότητα. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω το γεγονός ότι για λόγους συγκεκριμένους, επειδή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι, θα πρέπει και το Διευθύνσιο Προσματικό Ταμείο να συμμετέχει στη διαδικασία. Από κοινού με την Ευρωζώνη να γίνουν προσπάθειες δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχουν και οι νομικές, ε, τα νομικά κολλήματα. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε μαζί την Ελλάδα να φτάσει σε μια λύση αλλά θα ήθελα όλα αυτά να γίνονται μέσα στο πλέγμα κανόνων του ευρώ, της ζώνης του ευρώ, με τη συνδρομή του Διεθνούς Ταμείου, αλλά όχι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωζώνη. Ευρωζώνη με την αρρωγή του Διεθνούς Ταμείου. Αυτό ναι. Ό,τι μπορεί συμπληρωματικά δηλαδή να προσφέρει το δουνού του. Για την κυρία Λούλη. Θέσατε πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα να απαντήσω ότι αποκλείω την χρήση δανείων με την εγγύηση κρατών μελών ως πιθανό μέσον λύσης. Γιατί ένα, δύο ή και τρία ενδεχομένω κράτη της ζώνης ευρώ θα θέλαν να αποκλείσουν ένα κοινοτικό μέσον να το πω έτσι. Αυτή τη στάση θα μπορούσα και να τη σχολιάσω, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Με βλέπετε. Βλέπετε το πρόσωπό μου και την έκφρασή μου για να καταλάβετε τι σκέφτομαι στην πραγματικότητα για αυτή την υπόθεση. Άρα, αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε θα ήταν μια διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ των μελών της ζώνης του ευρώ που θα σήμαινε διάθεση στην Ελλάδα διμερών βοηθειών γιατί είναι το μόνο μέσο που έχουμε στη θέση μας. Εφόσον ε, αποκλείσουμε την περίπτωση των δανείων και έτσι σε αυτό θα έδινα την προτίμησή μου. Λέγοντα όμω ότι και πάλι δεν πιστεύω ότι πρέπει αμέσω να καταφύγουμε, γιατί είναι επαρκή οι προβλέψει και το πρόγραμμα τη Ελλάδα. Ε, πρόεδρε, επιτρέψτε μου, ε, εάν ο κάθε ένα από του ομιλητέ καταθέτει μία ερώτηση και όχι τρει, θα είναι πιο εύκολο να τελειώνω και εγώ την ε, απάντησή μου. Εσεί μιλήσατε για την κυρία Λαγκάρντ, επίση κυρία Λούλινγκ, ε, μια πρόσφατη τη δήλωση. Ναι, αλλά αυτή μην την αναμειγνύεται με το πρόβλημα τη Ελλάδα. Πρόκειται για μια δήλωση η οποία έχει να κάνει με μια άλλη κατηγορία προβλημάτων, τα οποία επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζώνη του ευρώ. Τις εσωτερικές δηλαδή ε, Ανισότητε ή αναισορπίε στην ε, ζώνη του Ευρώπη. Αλλά δεν επρώ τι προτεραιότητε αυτό το πρόβλημα πρώτα. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, γιατί τώρα έχουμε να λύσουμε το πρόγραμμα τη Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, οι συνολικέ, οι μάλλον εσωτερικέ ανισορποίηση ενισοπία, Η ανισορροπίε στην ζωνη του ευρω αλλα δεν ειναι πρωτη προτεραιοτητα αυτο το προβλημα πρωτον στην κατασταση που βρισκομαστε τωρα γιατι τωρα εχουμε να λυσουμε το προβλημα τη ελλαδα πρωτα απ ολα δευτερον οι συνολικε οι οποία οφείλεται στο γεγονό ότι ε, η Γερμανία έχει περισσότερο εχει περισσοτερη οταση προ τι εξαγωγέ και είναι ο κύριο κινητήριο. η κινητήρια δύναμη τη οικονομίας τη οι εξαγωγές δεν είναι ο μοναδικό λόγο αυτή τη ανισορροπία με στη ζώνη του ευρώ. Υπάρχουν άλλοι λόγοι και ευρύτεροι και πολύ πιο επικίνδυνοι. Απλώς θα θέλω να επισημάνω ότι τα κράτη-μέλη της ζώνης ευρώ που έχουν χάσει από την ανταγωνιστικότητά τους και έχουν σημαντικές διαρθρωτικές και χρόνιες ε, δυσκολίε και προβλήματα ανταγωνιστικότητας Πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστικότητά τους για να τη βελτιώσουν και μετά να κοιτάξουν το τι πρόβλημα γεννά η Γερμανία. Φυσικά αποδεχόμενος βέβαια το γεγονός ότι και η θέση και ο ρόλος της Γερμανίας είναι σημαντικός και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, πρέπει να το κοιτάξουμε το πρόβλημα αυτό. Επίση θα συμφωνήσω μαζί σας στην παρατήρηση ότι άλλα μεγαλύτερα από την Ελλάδα κράτη βλέπουν επιτέλους ότι ε, το να μην τηρεί κανείς τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη έχει συνέπειες ναι, αλλά ήμασταν πιο χαλαροί στην αντιμετώπιση κάποιων διολυστήσεων που είχαμε στο παρελθόν απέναντι στα κράτη αυτά, διότι υπήρχαν και διαφορετικές συγκυρίες και διαφορετικές σχέσεις ως προς και τα όμορα των μεγαλύτερων αυτών κρατών κράτη-μέλη. Και άρα μπορούσαν με κάποιες αρθρωτικές αλλαγές ε, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα πιο εύκολα. Το έλλειμμα βεβαίως είναι πολύ κατεπήγον πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα. Το έλλειμμα στο εξωτικό που ανέφερε η κυρία Νετφέλντ είναι κατεπήγον να αντιμετωπιστεί. Έχουμε γυράσκοντα πληθυσμό και στα προσεχή χρόνια αναμένουμε μεγάλους κλειδονισμούς που εάν δεν θεσπίσουμε συστήματα χρηματοδότησης πιο ουσιαστικά και πιο αξιόπιστα θα οδηγήσει σε κατάρρευση στα συστήματα της ταξιδότησής μας. Η χρηματοδότηση του συνταξιδοτικού μας συστήματος, του συστήματος γύρατος αν θέλετε, είναι ένα πρόβλημα σοβαρό, ένα πρόβλημα το οποίο θα επιτρέψει και στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και σε, άλλες, σε άλλους φορείς να κρίνουν, να αξιολογήσουν τις πολιτικές μας ως ικανοποιητικές σημεί. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρωζώνη να αποδείξει σε όλο τον πλανήτη, αλλά πάνω απ' όλα στους νέους που θα είναι εκείνοι που, θα, που καλούνται να ξεπληρώσουν τα χρέη μας, τα χρέη αυτών των στρατιωτικών μας συστημάτων, να αποδείξει ότι όλα μας τα συστήματα και όλα μας τα στραπογράμματα είναι αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα. Έχουμε να κάνουμε με ένα, πρόγραμμα, ένα πρόβλημα ε, αξιοπιστίας της παλιότερης γενιάς έναντι των νεωτέρων. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε νέο μιλητέ, λέει η πρόεδρο. 45 δευτερόλεπτο καθένα και θα σα κόβω γιατί αλλιώ δεν θα υπάρξουν απαντήσει. Έτσι και αλλιώ στις 25 θα σας κόψω όλους γιατί θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιούγκερ και πάλι. Θα σας πω ποιοι είσαστε. Roddy Kratzer, Robert Goebbels, Philippe Lambert, Annie Podimata, Pavanche Beres, Marian Tyson and Ramon Tremosa. So 45 seconds. 45 δευτερόλεπτα ο καθένας. President, mir scheint die Krise hat uns gelehrt. Κύριος Κλίντς, Έχω την εντύπωση, Πρόεδρε, ότι το πρόβλημα αυτό, η μεγάλη οικονομική κρίση δείχνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιστορική αγορά εκεί όπου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια μεγάλη φορολογική οικονομική ε, αγορά, εσωτερική αγορά. Όχι λιγότερη Ευρώπη, αλλά περισσότερη Ευρώπη δηλαδή. Τι λέτε εσείς. Ευχαριστούμε κυρία Ντατή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κρίση που περνάει η Ελλάδα σήμερα μας υποχρεώνει να έχουμε μια συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο οικονομική πολιτική. Αυτό είναι το βασικό. Την προηγούμενη εβδομάδα εσείς μαζέψατε τους ε, Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης για να μιλήσετε για την τεχνική πλευρά των ενισχύσεων για την Ελλάδα. Είμαστε ενωμένοι λοιπόν και για το καλύτερο και για το χειρότερο στην Ευρώπη. Σήμερα δεν μπορούμε εμείς ε, να είμαστε πια τόσο απαιτητικοί στην Ελλάδα για τα θέματα λιτότητος. Λοιπόν, εσείς είπατε ότι αν χρειαστεί βοήθεια θα δοθεί. Είπατε διμερής ε, βοήθεια από τη μια και από την άλλη Διεθνές ε, Νομισματικό Ταμείο. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς κύριε Πρόεδρε, ποια κατεύθυνση πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη. Έχετε κανένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη βοήθεια προς την Ελλάδα διακοπή της κυρίας Δατή. Λυπάμαι. Μα τελειώνω, λέει η κυρία Ντατή. Θέλω να μου πείτε πώς αντιδράτε στα όσα λέει η κυρία Μέρκελ για το Ευρωγκρουπ και στην αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία. Κόβει πάλι η πρόεδρος το μικρόφωνο της κυρίας Ντατή. Λυπάμαι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι, λέει η πρόεδρος. Δεν είναι δυνατόν. Θα κοπεί ο επόμενος και μετά δεν θα ακούσουμε κανέναν άλλον πια. Η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχομαι στο θέμα της Ελλάδας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργό έχει κάνει πολλά και σαφές ότι δεν ζητά οικονομική υποστήριξη, δεν ζητάει χρήματα. Το επαναλάβατε και εσείς σήμερα. Τι ζητάει η Ελλάδα? Ένα μήνυμα σαφές στις αγορές για να αρχίσουν να πέφτουν τα επιτόκια δανεισμού. Αυτό όμως το μήνυμα το έχει ανάγκη άμεσα διότι η Ελλάδα έχει άμεσα ανάγκη δανεισμού. Τα μέτρα μέχρι τώρα δεν έχουν πείσει τις αγορές. Όχι τα, η κατάσταση ελληνική, ε, το ελληνικό πρόγραμμα και η κοινοτική βοήθεια. Πώς πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να είναι αυτή η βοήθεια, ώστε να θεωρηθεί επαρκής για τις αγορές. Η εκατέρωθεν προσπάθεια πώς μπορεί να είναι επαρκής. Και το θέμα είναι άμεσο, δεν είναι όταν το χρειαστεί η Ελλάδα. Euh, Ευχαριστώ. Σε κάθε νομισματική ζώνη οι σχέσεις εξορισμού είναι ασυμμετρικές. Κάποιοι έχουν παραπάνω έλλειμμα, κάποιοι λιγότερο. Αυτό ισχύει και στι Ηνωμένε Πολιτείε και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρε καλύτερε, με καλύτερε επιδόσει από ό,τι άλλε. Εσεί αναφερθήκατε στην ε, Καλιφόρνια, που σίγουρα σε απόλυτου όρου είναι σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα. Λοιπόν, η... είναι γεγονό ότι και οι Κινέζοι χρηματοδοτούν σε ένα βαθμό την ε, Ευρώπη και το ρόλο των Κινέζων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον παίζουν οι Γερμανοί. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει προπολογισμό αντίστοιχο με τι ανάγκε. Αν μη τι άλλο, πρέπει να έχουμε μια εσωτερική αγορά για τα Eurobonds, τι ευρωμετοχέ, ώστε ο καθένα να μπορεί να, μπορεί να χρηματοδοτείται εκ νέου. Είναι φίλοι. Ευχαριστώ κύριε Γιούνκερ. Καλώ ήρθατε στι Βρυξέλλε. Είναι απλή η ερώτησή μου. Φυσικά και πρέπει να λύσουμε αυτή την εξίσωση τη δημοσιονομική και να επανέλθουμε σε πιο υγιή ευρωπαϊκά δημοσιονομικά. Πώ θα το κάνουμε αυτό, μόνο κοιτώντα τι δαπάνε και χωρί να κοιτάμε τα έσοδα. Ρωτάω λοιπόν, πόσο καιρό μπορούμε να συνεχίσουμε να μην έχουμε φορολογική σύγκληση. Το κάνουμε για το ΦΠΑ, γιατί όχι και για τα υπόλοιπα. Άννη Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ <clears throat> και εσάς. Είσαστε εξαιρετικά σαφείς στις απαντήσεις σας σε σχέση με έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό υποστήριξης της Ελλάδας. Εφόσον χρειαστεί υπογραμμίσατε, εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι σημαίνει εφόσον χρειαστεί, διότι εφόσον χρειαστεί είπαμε και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 Φεβρουαρίου ε, η Ελλάδα ξαναβγήκε στις αγορές στις 5 Μαρτίου και δανείστηκε με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δανειστεί με επιτόκια παρεμφερή με αυτά που υπήρξαν στις 5 Μαρτίου. Το ερώτημα λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεθαύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ελλάδα αναγκαστεί να καταφύγει σε άλλες λύσεις εκτός Ευρώπης για να εξασφαλίσει χαμηλά επιτόκια δανεισμού ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για το ευρώ και για την ευρωζώνη συνολικά. Μία παρατήρηση. Εγώ σοκαρίστηκα όταν το τελευταίο συμβούλιο εκοφήνε πήρε την απόφαση για την απόσυρση των μέτρων για την αγορά εργασίας. Λοιπόν, για την Ελλάδα, από τον Οκτώβριο του 2008 ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και πολλοί είχαν πει τότε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 122 για να αντιμετωπίσουμε την ελληνική κρίση. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε πάλι για το σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο λειτουργεί ακόμη πιο κατασταλτικά. Τελικά ο ρόλος του δεν είναι η όξυνση των ανισοτήτων παραγωγικότητας μεταξύ κρατών μελών. Δεν χρειαζόμαστε ένα σκληρό μέσο, ένα πιο απαλό μέσο χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κυρίος Χωσέ Μαριολάντα από την, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, από την Ισπανική Τράπεζα είπε ότι ο τομέας των ακινήτων στην Ισπανία με 150.000 ευρώ που είναι το 45% του ΑΕΠ και επίσης ο κύριος Ναβάρο που είναι πρόεδρος ε, του Ισπανικού Επιμελητηρίου είπε ότι 30% του ποσού αυτού δεν θα ε, ανακτηθεί ποτέ. Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα για το ευρώ. Um, Κύριε Γιούνκερ, στις 5 έχουμε τον κύριο Τρισέ, οπότε Α, άρα έχω καιρό. Τέσσερα μισή, τεσσεράμιση τέσσερα είναι ο κύριος Τρισέ. Ας μπει όμως, ας περάσει, ας έρθει, ας καθίσει. Ας το ανοίξει κάποιος την πόρτα. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, διότι σε ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις είτε έχω απαντήσει εξ ολοκλήρου, είτε μερικός. Οπότε δεν θα τα ξαναπώ. Για την Ελλάδα ήθελα να πω, γιατί πολλές ερωτήσεις στράφηκαν σε θέματα που ανέφερα. Πρώτον λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης του προϋπολογισμού της και εξηγία της των των δημοσιονομικών της. Δεύτερον, η Ελλάδα, τόσο η κυβέρνηση όσο και το κοινοβούλιο ενέκριναν μέτρα εντελώς αξιόπιστα τα οποία δείχνουν ότι η βούληση της Ελλάδας είναι να κερδίσει το στοίχημα. Τρίτο, αν συνεχιστεί η σπέκουλα, η κερδοσκοπία των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι της Ελλάδος, ενώ η Ελλάδα έχει κάνει τα πάντα για να εξηγιάνει τα οικονομικά της, η Ευρωζώνη πρέπει να είναι έτοιμη και θα είναι έτοιμη για να βοηθήσει την Ελλάδα βάσει ενός μέσου το οποίο δεν θα σας το αποκαλύψω σήμερα στις λεπτομέρειές του αλλά το οποίο θα το έχουμε στη διάθεσή μας όταν έρθει η ώρα. Τέταρτον, όλη η ιδέα αποκλεισμού μίας χώρας από την Ευρωζώνη νομίζω ότι είναι μία ιδέα παράλογη. Κανένας δεν πρότεινε να αποκλειστεί η Ελλάδα, να αποβληθεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Όλες οι συζητήσεις που έγιναν προς αυτήν την κατεύθυνση δεν αφορούσαν στην ελληνική περίπτωση, αλλά σε ένα μέσο που θα έπρεπε να πρικοδοτηθεί ίσως η Ευρωζώνη κάποτε ή η Ένωση για το μέλλον. Ο παραλληλισμός ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι ούτε εντελώς αληθινές ούτε εντελώς ε, στρεβλές. Αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια χώρα με κεντρική εξουσία, με αρμοδιότητες κεντρικές. Η Ευρώπη δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Δεν έχει δηλαδή τα μέσα που μπορούν οι κεντρικές κυβερνήσεις ε, να ενεργοποιήσουν. Έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξη. Εντάξει, μπροστά στο Λότελα, καλό είναι και αυτό. Αλλά Ε, λέω σε εσά λοιπόν κυριέ μου ότι ναι χρειάζεται ένα μήνυμο με ε, για τα φορολογικά. Το κάναμε το 91 για τον ΦΠΑ και τα τέλη και τους δασμούς. Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε και για άλλα θέματα φορολογικού χαρακτήρα. Χωρίς βέβαια να καταργήσουμε την, τον υγιή ανταγωνισμό που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ κρατών μελών της ίδιας ζω, ε, ζώνης. Λοιπόν, εγώ είχα μιλήσει για τα Eurobonds, για τα ευρωμόλογα πριν από μερικά χρόνια, τρία χρόνια έχει η Ρομπέχ και δεν ε, συμφώνησαν. Θα είχα πολλές ευκαιρίες να το θυμίσω αυτό στους συνομιλητές μου τότε ε, ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν με ακούσανε. Ε, λοιπόν, ε, τώρα χρειάζεται να, ίσως να προσφύγουμε στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν ναι ή όχι, τέλο πάντων χρειάζεται τροποποίηση των συνθήκων ή μπορεί να βρεθεί μια λύση αυτού του στυλ μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που έχουμε είναι άκυρη η συζήτηση σήμερα, αλλά την επόμενη φορά θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ένα μέσο το οποίο να το δραστηριοποιήσουμε χωρίς ιδιαίτερα δράματα και χωρίς ε, αμφισβητήσεις αρχών όπως γίνεται σήμερα. Χρειάζεται να πω ότι ναι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά ούτως ώστε το οικοδόμημά μας να είναι πιο, πιο γερό και πιο συνεκτικό. Εγώ πάντα έλεγα ότι το άρθρο 122 της συνθήκης δεν είναι νομική βάση της προκοπής όπου μπορούμε να βαθισίσουμε οποιαδήποτε δράση υπέρ της Ελλάδας. Εγώ λοιπόν θα έλεγα στην κυρία Ντατή ότι ναι, μπορώ να την ακολουθήσω στη σκέψη της ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την εξυγίανση των οικονομικών της, αλλά και οι χώρες της Ευρωμάδας πρέπει να είναι έτοιμες να επικουρήσουν την Ελλάδα, να τη βοηθήσουν αν η Ελλάδα χρειαστεί οικονομική υποστήριξη από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η ιδέα τώρα για να αποκλείσουμε, να αποβάλουμε μια χώρα από τη ζώνη ευρώ το είπα και πριν και το ξαναλέω ότι είμαι αντίθετος και αν θέλουμε εμείς έναν μηχανισμό που να αποκλείει, να αποβάλει ένα κράτος μέλος, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ένας μηχανισμός όπου ο καθένας να μπορεί να φεύγει και κατά τη βούλησή του. Αυτό φυσικά θα αποσταθεροποιούσε την ε, νομισματική ζώνη στο σύνολό της. Λοιπόν, εγώ σέβομαι την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, γι' αυτό λοιπόν θα τελειώνω στο Pix Lux. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που συσσωρεύσαμε τόσο πολλές ερωτήσεις και σας δυσκολεύσαμε τόσο πολύ στο έργο σας. Ελπίζω ότι στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε προβλέψει για τις 4 Οκτωβρίου να σας ξαναδούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Ζήνκερ. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, 2-3 λεπτών. Okay, everybody, if you could uh, sit. Παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε και πάλι. Είναι δύσκολο κάθε φορά που έχουμε τόσο εξέχοντες προσκεκλημένους. Τώρα λοιπόν καλωσορίζω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Έρχεται κάθε τόσο, έχουμε τακτικά διάλογο μαζί του και περιμένουμε και πάλι να μας μιλήσει και για την Ελλάδα, μια που είναι ένα θέμα που μας ε, απασχολεί. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξει σίγουρα. Ο κύριος Τρισέ, 15 λεπτά περίπου, θα κάνει την παρουσίασή του και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις όπως κάνουμε συνήθως. Έχω εδώ όσους έχουν ζητήσει να υποβάλουν ερωτήσεις. Πάντως, παρακαλώ, μην υποβάλλετε πολλές και περίπλοκες ερωτήσεις με μιας. Γιατί έτσι δεν προλαβαίνουν οι υπόλοιποι και είναι πολύ δύσκολο και ο κύριος Τρισέ να απαντήσει τότε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Τρισέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και σας δίνω το λόγο ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα για την πρώτη αυτή συνάντησή μας για το 2010. Τους τελευταίους μήνες μετά την τελευταία μας συνάντηση το Δεκέμβριο του 2009, ο ευρωχώρος και η οικονομία του ευρωχώρου στο σύνολό της άρχισε ανάκαμψη. Όμω παραμένουν θέματα που έχουν να κάνουν με διάφορε χώρε ή με τι εξελίξει στι δημοσιονομικέ αγορέ που οδήγησαν σε έντονε συζητήσει για τον ευρωχώρο και για τη λειτουργία του. Έτσι η σημερινή μα συζήτηση είναι πάρα πολύ επίκαιρη βλέπουμε ποιες είναι οι μεγάλες ε, προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν ε, ως ε, προκλήσεις για την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική μάλλον κρίση. Και βλέπουμε τι σημαίνει το να αντιμετωπίζει κανείς με υπευθυνότητα την ε, οικονομική και νομισματική πολιτική. Η σταθερότητα του κοινωνομίσματος είναι ευθύνη όλων μας. Σήμερα, όσοι ήθιστε, θα ξεκινήσω με μια αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην σταδιακή κατάργηση των ε, έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν κατά την περίοδο της κρίσης. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στα δύο θέματα για τα οποία έχουμε συμφωνήσει, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική και τις ε, ανισορροπίες παγκοσμίω. Πρώτα απ' όλα για τι οικονομικέ και νομισματικέ εξελίξει. Όπω είπαμε, από το Δεκέμβριο που μα πέρασε, οι οικονομικέ και δημοσιονομικέ συνθήκε έχουν βελτιωθεί σε έναν μέτριο βαθμό. Η οικονομική δραστηριότητα έχει αυξηθεί κατά 0,1% το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Και οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε λένε ότι περιμένουμε επίσης μία συνέχιση της ανάκαμψης τα επόμενα, το υπόλοιπο της χρονιάς. Όλα αυτά βέβαια συνάδουν με τις αξιολογήσεις και τις εκτιμήσεις που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε ένα μέσο ε, ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης 1% το 2010 και θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί το 2011. Στην ε, εκτίμηση και την αξιολόγηση που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι κίνδυνοι ε, είναι σε μεγαλύτερη ισορροπία τώρα και προβλέπεται, όπως είχαμε ήδη προβλέψει και από πέρυσι, ανάκαμψη που όμως δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις χώρες. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις στις τιμές, έχουμε συνεχίσει να διαπιστώνουμε χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις τους πρόσφατους μήνες. Το Φεβρουάριο του 2010 ήταν 0,9%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει ε, σε αυτά τα επίπεδα με τη σταθερότητα των τιμών, μια που οι κίνδυνοι παραμένουν σε ισορροπία. Περιμένουμε ο πληθωρισμός να παραμείνει στο 1% εξαιτίας της χαμηλής ανάκαμψης στη ζήτηση. Η νομισματική μας ανάλυση εξακολουθεί να επιβεβαιώνει τις προοπτικές για χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, όπως φαίνεται από την χαμηλή ανάπτυξη της τιμής του χρήματος και των πιστώσεων. Η αύξηση των δανείων παραμένει χαμηλή, ενώ η, ανάπτυξη, μάλλον ενώ η αύξηση των επιτοκίων των δανείων για τα νοικοκυριά ε, ενισχύεται. Αυτές ε, βέβαια εξελίξεις συνάδουν με την επανάληψη των κύκλων όπως γνωρίζουμε. Εμείς θα παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει περιορισμός ε, των πιστώσεων στην ε, Ευρωζώνη. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια και από τις επιχειρήσεις, από το μέγεθός τους κλπ. Πάντως, η χαμηλή ανάπτυξη όσον αφορά τα δάνεια οφείλεται στην πολύ σοβαρή ύφεση που είχαμε το 2009. Οι δείκτες πάντως για τις προπτικές στον πληθωρισμό, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, παραμένουν σύμφωνα με τους ε, στόχους κοντά στο 2% θέλουμε μεσοπρόθεσμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, κράτησε ε, σταθερά τα επιτόκια. Αυτό αποφάσισε πριν από ένα μήνα περίπου. Η σημαντική τώρα νομισματική όθηση είναι απόρρια των χαμηλών επιτοκίων πέρυσι και αντικατοπτρίστηκε και στα επιτόκια στις αγορές και στη συνέχεια ε, στα επιτόκια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Η πρόβλεψη για ρευστό στις τράπεζες για ένα διάστημα ενός χρόνου για να αποφύγουμε τους κινδύνους έφερε αποτελέσματα και έδωσε στις τράπεζες ευνοϊκές συνθήκες ώστε να σταθεροποιηθεί η νομισματική αγορά και να ενισχυθεί η μείωση των επιτοκίων μας. Τώρα, βάσει των αξιολογήσεων αυτών, των οικονομικών και των νομισματικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε στις αρχές του μήνα να συνεχίσει να μειώνει τα έκτακτα μέτρα. Δεν θέλουμε εμείς να καλλιεργήσουμε την εξάρτηση από τέτοια μέτρα. Οι τράπεζες, η τράπεζα ε, θέλει να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να πάψουν αυτά τα εκτακτά μέτρα. Έτσι κι έχουν σταματήσει οι δωδεκάμενες επιχειρήσεις και η εξάμηνη τελευταία θα σταματήσει την επόμενη εβδομάδα. Επιπλέον σκοπεύουμε να προσφέρουμε ε, μεταβλητά επιτόκια στις τρίμηνες επιχειρήσεις μας στα τέλη του Απριλίου. Συγχρόνως θέλουμε το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης να έχει απεριόριστη πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα μέσω βραχυπρόθεσμων ε, δράσεων όσο χρειαστεί αυτό και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου της χρονιάς αυτής. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε λοιπόν την οικονομία της Ευρωζώνης με τέτοιες πιστώσεις. Τώρα επιτρέψτε μου να πω και μερικά πράγματα για την μακροπρόθεσμη νομισματική μας πολιτική που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, ιδιαίτερα σε σχέση με την νομισματική πολιτική και την τιμή των ακινήτων. Η δημοσιονομική κρίση ξανάδειξε ότι υπάρχει θέμα στη σχέση ανάμεσα στην νομισματική πολιτική μας και τις φούσκες από τις τιμές των ακινήτων. Η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με το εξή ζήτημα. Πρέπει η εποπτική μας πολιτική να αποφεύγει τη δημιουργία τέτοιων ε, κρίσεων όπως ε, μετακίνητα. Ε, το θέμα βέβαια δεν έχει μια απλή απάντηση. Πάντως η δική μας νομισματική πολιτική και στρατηγική είναι να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που δημιουργούνται από μη βιώσιμες εξελίξεις στην τιμή των ακινήτων εντολή μας είναι να διατηρούμε την σταθερότητα τιμών μεσοπρόθεσμα ε, συνεχώς και οι διάφορες ε, αυξομοιώσεις στις τιμές των ακινήτων σίγουρα δημιουργούν κινδύνους όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών. Η σχέση ανάμεσα στις νομισματικές εξελίξεις και στις ανισορροπίες που υπάρχουν στα κίνητα και στις πιστοτικές ε, αγορές επιβάλλουν αντιμετώπιση σε πρώιμο στάδιο και μια απάντηση για να αποφεύγονται κίνδυνοι από την αστάθεια τιμών. Προκειμένου βέβαια όλα αυτά για να έχουμε ε, δημοσιονομική σταθερότητα. Η νομισματική μας ανάλυση που επικεντρώνεται στην εποπτεία των ε, θεμάτων αυτών είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε σε ένα βαθμό ε, άρρητα παρέμβαση από την πλευρά μας, αυτό που λέμε leaning against the wind, για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Φυσικά πάντα πρέπει να κρίνεται η κατάσταση ανάμεσα με το τι δυνάμει περιμένουμε. Πάντως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εμπειρία σε αυτά τα θέματα, αναλύει λοιπόν την κατάσταση όσον αφορά τις νομισματικές και τις πιστοτικές ε, εξελίξεις και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη σταθερότητα τιμών. Τώρα θα έρθω λίγο στη δημοσιονομική πολιτική. Όπως ξέρετε, ε, τα τελευταία γεγονότα, στήριξη του δημοσιονομικού τομέα, όπως επίσης και η χαλάρωση των δημοσιονομικών, οδήγησαν σε ανισορροπίες. Συγχρόνως, πολλές χώρες στην Ευρωζώνη έχουν ξεπεράσει τον αριθμό αναφορά στο 3% δηλαδή για το έλλειμμά τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που φροντίζει για η υγιή δημοσιονομικά πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν ζητάει να ε, ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο η δέσμευση των κυβερνήσεων υπέρ της στήριξης των όρων του συμφώνου αυτού. Η εθνική πολιτική πρέπει να δώσει αυτό το θέμα μεγάλη προτεραιότητα ώστε να επανέλθει το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ όπως λένε και οι συστάσεις οι πρόσφατες του ΕΚΟΦΗΝ. Βάσει του προγράμματος σταθερότητας οι κυβερνήσεις φαίνεται να προχωράνε προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά αναμφίβολα θα χρειαστούν και άλλα μέτρα τις επόμενες χρονιές προκειμένου να αποφύγουμε υπερβολικά ελλείμματα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τώρα την σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής, χαιρόμαστε που περιορίζονται οι δαπάνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο δημόσιος τομέας έχει επεκταθεί πολύ και έχει συνεισφέρει αυτό στην κρίση ενώ πρέπει η εξυγίανση των δημοσιονομικών να βοηθήσει στη συνέχεια. Οι κυβερνήσεις πρέπει να φροντίσουν να ενισχύσουν ε, τα μέτρα τους για δημοσιονομική ρύθμιση και να εφαρμόσουν διευθυντικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Οπότε χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στρατηγική Ευρώπη 2020 και για τον ενισχυμένο ρόλο του Eurogroup στην ε, πολυμερή εποπτεία χωρών. Συγχρόνως είναι σημαντικό η δημοσιονομική εποπτεία βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας να παραμείνει μια ε, διαδικασία αυτοδικαίως και να τηρούνται οι διατάξεις της συνθήκης και του Συμφώνου πλήρως. Για να βγούμε από την κρίση χρειάζονται, χρειάζεται περιορισμό των υψηλών δημοσιονομικών δαπανών. Οι υπεύθυνοι πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν να επανέλθει το σύστημα σε ανεγές επίπεδο και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί πρόσφατα από την Ιρλανδική κυβέρνηση και ακόμα πιο πρόσφατα από την ελληνική κυβέρνηση αποτελούν πολλά υποσχόμενα πρώτα στην επερχόμενη διαδικασία εξυγένσης. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και για τις ανισορροπίες. Ένας από τους κύριους λόγους που μας οδήγησε στην οικονομική κρίση ήταν ε, ακριβώς οι εξωτερικές αυτές ανισορροπίες, που είχαν σαν αποτέλεσμα μαζικές ροές κεφαλαίων σε χώρες με λύματα. Αυτές οι ροές χρηματοδοτήθηκαν σε ένα βαθμό από δημοσιονομικά ε, μέσα, τα οποία συνεισέφεραν στι ανισορροπίε αυτές, οι οποίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει μεσοπρόθεσμα σωστό προσανατολισμό υπέρ τη σταθερότητα και της βιωσιμότητα της μακροοικονομικής πολιτικής σε χώρες είτε ελληματικέ είτε πλεονασματικές. Ο ευρωχώρος δεν συνεισέφερε στην οικοδόμηση των ανισορροπιών αυτών. Όχι. Η ισορροπία παρέμεινε σχετικά τα τελευταία χρόνια. Η κρίση οδήγησε σε μία μείωση τελικά των ε, ανισορροπιών, αλλά η διόρθωση αυτή βασίζεται σε κύκλους. Υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν ε, σε ανισορροπίες και παραμένουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποκλείσουμε στην επόμενη περίοδο που έχουμε μπροστά μας ξανά τέτοιου είδους ανισορροπίες. Για να τις αποφύγουμε χρειάζεται προσαρμογή με λιτότητα για να αποφύγουμε νέα ελλείμματα. Η απόφαση των 20 να δημιουργήσουν μια διαδικασία για μακροοικονομική και διευθυντική πολιτική και μια αμοιβαία ε, αξιολόγησή της καθετόσο είναι θετική. Χρειάζεται όντως εποπτεία από μότυπους προκειμένου να μπορέσουμε χωρίς ε, υποχωρήσεις και δίκαια να ελέγξουμε τις χώρες και τις οικονομίες ε, που πρέπει να αλλάξει η εσωτερική πολιτική των χωρών αυτών σύμφωνα με τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι ο Ευρωχώρος μπορεί με θετικό τρόπο να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να πετύχει τη σωστή μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ε, πολιτική. Θα ολοκληρώσω με το εξή. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες υπάρχουν και μέσα στην Ευρωχώρα, δεν είναι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν μια πρόκληση η οποία δείχνει ότι λείπει η προσαρμογή σε πολλές χώρες μέλη. Είναι αναγκαίο λοιπόν οι χώρες αυτές να φροντίσουν για να ελέγξουν τους δείκτες της ανταγωνιστικότητάς τους και να διορθώσουν με μεταρρυθμίσεις ότι χρειάζεται για να πετύχουν εξυγίαση των δημοσιονομικών τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης να υποφεληθούν πλήρως από την Οικονομική και Νοσματική Ένωση. Uh, uh, Σας ευχαριστώ. συνήθως οι ερωτήσεις θα έχουν περιθώριο 1,5 λεπτό, οι απαντήσεις 3 λεπτά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το διάλογο. Ο Ζων Πολγκοζέσης πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω, όπως και στον κύριο Γιούνκερ, ότι οι συμπολίτε μας ε, δεν καταλαβαίνουν πια τι συμβαίνει εν γέννη έχουν εμπιστοσύνη στο ευρώ, εν γέννη έχουν καλή εικόνα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέσα στους σημερινούς κλειδονισμούς όμως δεν αντιλαμβάνονται πλέον εάν βρισκόμαστε μέσα σε μια ζώνη αλληλεγγύης με ένα κοινό νόμισμα, με ένα ενιαίο νόμισμα ή εάν υπάρχουν πάλι αντιπαραθέσεις και διελκυστίνδες των μεν εναντίον των δε ως προς το με ποιο τρόπο ε, συμπεριφερόμαστε απέναντι στα μέλη της Ευρωζώνης. Η θέση σας και την εκτιμώ ιδιαίτερως, θέση που υιοθετήσετε δημοσία και θα ήθελα να ζητήσω να επανέλθετε ως προς το τι θεωρείτε ακριβώς αποδεκτή ε, βοήθεια προς την Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο πράγμα τη δυσκολίες. Θα σαφείς λοιπόν θέσεις και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω, μια δεύτερη ερώτηση, εάν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο ή όχι, ή τόσο τι θεωρείτε, ως προς το εάν χρειάζεται να ενισχυθεί η προληπτική πτυχή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που εμφανίζονται με κάποιες καθυστερήσεις ενδεχομένω δυσκολίες σε ένα κράτος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Τρισέ, για την ερώτηση σα. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και να πω καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντοτε απέδιδε τη μέγιστη σημασία στην δημοσιονομική φρόνηση. Το έχουμε αποδείξει αυτό άλλωστε και σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί στην περίοδο 2004-2005 τα περισσότερα κράτη-μέλη θέλανε να απαλλαγούν από το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Και εγώ ήμουν εκείνο, πρέπει να σα επισημάνω, ότι τρία, τα τρία μεγαλύτερα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ζώνη, όπω του Ευρώπη τότε, θεωρούσαν ότι θα πρέπει να ε, το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Τέλο πάντων, η επιπτώση του. Εμεί όχι, υπεραμεινθήκαμε αυτού με σθένο και είπαμε: Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι τρία γράμματα. Όμικρον, νη, έψιλον. Εμείς έχουμε το νη, την νομισματική ένωση, αλλά χρειαζόμαστε το όμικρον, την οικονομική και αυτό σημαίνει δημοσιονομική φρόνηση και επίση επιτήρηση από του ομοίου, από του ομολόγου Αυτό το να, επιτηρεί, να επιτηρούν οι ομόλογοι οι εταίροι, αυτό που κάνει ο εταίρος, είναι και το καλύτερο μέσον ελέγχου. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς ε, να αποδεικνύεται περίτρανα αυτό που είπαμε ανέκαθεν ότι εάν παραμεληθεί η δημοσιονομική φρόνηση ως παράγον τη νομισματική πολιτική έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα. Και συμφωνώ απολύτω σε αυτό το οποίο είπατε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια το, το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη το οποίο εφευρέθηκε ακριβώ για να ενισχυθεί η προληπτική πτυχή και όχι για να αποδυναμωθεί η πτυχή των κυρώσεων. Αυτό το Σύμφωνο λοιπόν σταθερότητα και ανάπτυξη θα πρέπει με αυστηρότητα να τηρείται όπω πάντοτε. Στι υφιστάμενε τώρα συνθήκε. Θα σα πω τα εξή. Πρώτον, φρονώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε προσεκτικοί και αυστηροί στους όρους που χρησιμοποιούμε. Η πειθαρχία δηλαδή, η γλωσσική έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ακούγονται διαφορετικές δηλώσεις από διαφορετικά όργανα. Θα ήθελα και εγώ να κάτσουν κάτω μαζί τα θεσμικά όργανα, να συζητήσουν και να προσδιορίσουν από κοινού και με σαφείς όρους τις θέσεις τους. Όπως άλλωστε έγινε και στο τελευταίο, στην τελευταία σύνοδο κορυφής, όπου νομίζω ότι αρχικά των και κυβερνήσεων διατύπωσαν μια σαφή θέση και την οποία σαφώς και αντελήφθη η κοινή γνώμη, ο αποδέκτης πάνω απ' όλα των θέσεων αυτών την αντελήφθη και βέβαια όπως είδαμε ελήφθησαν και οι νέες αποφάσεις από την ελληνική κυβέρνηση όπως άλλωστε όλοι γνωρίζουμε μέσα σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Και για την τρίτη σας ερώτηση, δύο λόγια, τους όρους προσφοράς ενίσχυσης ή υποστήριξης. Φρονώ ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής όροι. Πρώτον, να μην μπερδεύουμε την μεταφορά ή την ε, επιδότηση με ένα δάνειο το οποίο θα είναι του τύπου θα είναι του τύπου αυτόν που δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. γιατί εδώ ακριβώς είναι η διαφορά. Με, τις, ε, με τη δική μας δυνατότητα παροχής βοήθειας. Επίσης, πέραν των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα πρέπει να υπάρχει μια αυστηρή πολιτική, άλλωστε το βλέπουμε αυτό με, τους, με τα νέα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης και εμείς οι ίδιοι τα χαρακτήρισαμε θαραλέα μέτρα και στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα χαρακτήρισαμε πιστικά μέτρα και είναι ένας από τους όρους αυτούς, αλλά αυτό δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με τα δάνεια του Δομιστικού Ταμείου που έχουν άλλου ίδιους εξαρτήσεις και ειδικού όρους. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πάλι για μία στήριξη όχι επιδοτικής φύσεως και όχι βάση ειδικών όρων, τύπου Διεθνούς Προστατικού Ταμείου, θα είναι πράγματι ένα κράτος να την χρειάζεται την ενίσχυση αυτή, δηλαδή να έχει βαρύτατα και άμεσα προβλήματα να αντιμετωπίσει, να μην είναι δηλαδή τρέχουσες υποθέσεις, αλλά έκτακτες περιστάσεις αυτές που το υποχρεώνουν να στην ενίσχυση. Και αυτές οι έκτακτες περιστάσεις θα πρέπει να προξενούν ζήτημα για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, όπως άλλωστε επεσήμεναν και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη δήλωσή τους. Αυτή είναι η όρη τους οποίους θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως απαραίτητους για τη χορήγηση μιας τέτοια ενίσχυσης όρου, Δηλαδή, όχι με ειδικού όρους, ε, συνθήκες δηλαδή δεσμευτικές, αλλά προϋποθέσεις συγκεκριμένες και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς το σύνολο της ζώνης του ευρώ, δηλαδή την δυνατότητα αποσταθεροποίησης, την πιθανότητα μάλλον αποσταθεροποίησης της ζώνης του ευρώ. Με συγχωρείτε Πρόεδρε που πακρηγόρησα, ξέρω ότι σας ε, προξενώ δυσκολίες και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ, προσπαθώ να, διατηρώ, να τηρώ και την πειθαρχία των συναδέλφων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τρισέ που ήρθε εδώ. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην παρατήρηση που κάνατε πριν για το προληπτικό σχέ... Ε, σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας. Είπατε ότι αυτό το προληπτικό σκέλος πρέπει να ενισχυθεί και ότι πρέπει να φροντίσουμε για την εφαρμογή του. Τώρα, η πρόσφατη ιστορία μας έχει δείξει ότι αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Η Γαλλία, η Γερμανία ε, έχουν φροντίσει νομίζω και σήμερα αν κοιτάξουμε τι παραδείγματα έχουμε όσον αφορά την εποπτεία των τραπεζών και αν λάβουμε υπόψη μας τους συμβασμούς τους οποίους κατέληξε το Συμβούλιο, του Συμβούλιο τους τόσο αδύναμους καταλαβαίνετε ότι η λύση δεν είναι κοντά. Το προληπτικό σκέλος λοιπόν είπατε πρέπει να ενισχυθεί. Ε, λοιπόν συγκεκριμένα πώς θα το κάνετε. Τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχυθεί αυτό το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει τα δημοσιονομικά των χωρών, να μην εξαρτάται από τα κράτη-μέλη μόνο το τι θα κάνουν ή έχετε κι άλλες προτάσεις. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε λοιπόν αυτό το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ερώτησή σας. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο που λέτε ότι κάποια στιγμή ακόμα και χώρες που δεν είναι τόσο συνηθισμένο να το ζητάνε καταλήγουν να ζητήσουν αποδυνάμωση. Τον Ιανουάριο λέγαμε η πολιτική μας μπορεί να οδηγήσει στην συμμόρφωση με το σύμφωνο σταθερότητας. Έχουμε τους σωστούς δείκτες. Όχι. Τα πιο σημαντικά κριτήρια θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση, που είναι η απασχόληση για παράδειγμα, Όλα αυτά ήταν αναγκαία και τα ζητήσαμε. Αλλά σίγουρα τα γνωρίσαμε στη συνέχεια. Μιλάω για το, την εκτελεστική πτυχή του ελέγχου. Πάντως εγώ πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα για να προλάβουμε τέτοια γεγονότα είναι κάθε μέλος της Ευρωζώνης και μιλάω μάλλον και για τους 27 διότι το σύμφωνο σταθερότητα επιβάλλει και στους 27 τα πράγματα. Αλλά στην Ευρωζώνη υπάρχουν κυρώσει, Αυτή είναι η διαφορά. Μπορούν να αποφασιστούν κυρώσει από τους πίεσε, από τους ε, ομότιμους ε, που αναλαμβάνουν την εποπτεία. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν για μένα το βασικό πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε τέτοιους ε, ομότιμους επόπτες οι οποίοι πιέζουν τις χώρες μέλη και κυρίως τα μέλη της Ευρωζώνης που δεν συμμορφώνονται. Τώρα έχουμε δει ότι οποιοδήποτε από εμά μπορεί να επηρεάσει την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Το έχουμε μπροστά μας, ζωντανό το παράδειγμα. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να ξυπνήσουμε και να αναλάβει κάθε κυβέρνηση ή χώρας μέλος τις ευθύνες της, ιδίως μέσα στην Ευρωζώνη. Συνεπώς, η χωρας μέλους τις ευθυνες της ιδιως μεσα στην ευρωζωνη συνεπως η αποφασιστικοτητα για να επιβάλλουμε, αν μη τι άλλο, ηθική πίεση, είναι μια πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα, όπως είπατε και εσείς, και σε άλλους τομείς. Να υπάρξει μεταφορά χρημάτων βάσει των συνήθων μηχανισμών. Καλά, πολλές, πολλά κανάλια μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι υψηλό επίπεδο ευθύνης του καθενός και πολιτική δέσμευση υπέρ της σταθερότητας. Πίεση από τον έλεγχο που κάνουν οι ομότιμοι. Αυτό είναι το βασικό. Ευχαριστώ κύριε Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Έρχομαι στο θέμα που αναφέρατε, ο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει την εξάρτηση από την υποστήριξη και τα έκτακτα μέτρα. Ε, και το εντάσσω στο, στην περίπτωση της Ελλάδας. Θα δεχόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελληνικά κρατικά ομόλογα με χαμηλότερη αξιολόγηση ως ενέχειρο για τα δάνεια που χορηγεί ως ένα μέσο συμπαράστασης στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει η ελληνική οικονομία και η προσπάθεια εξυγίανσης και ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. We accept as... Ναι. Ως ε, εγγύηση μπορούμε να πάρουμε τα... Βέβαια, τα ελληνικά ομόλογα μπορούμε να τα παίρνουμε. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. ενώ στην, ε, πορεία απόσυρσης των μέτρων υποστήριξης. θα έχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση Ελλάδα. Δεν λέω για σήμερα, το ξέρω ότι δέχεται. Αλλά στην πορεία που θα έχει η τράπεζα, αποσύροντας τα μέτρα ιδιαίτερης στήριξης, εάν σκέφτεστε να είναι προσφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μια ιδιαίτερη μεταχείριση προς την Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση, διότι θα ε, συνεχίσει να έχει ανάγκη μιας υποστήριξης περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες που έχουν λιγότερες συνέπειες της κρίσης. Σας ευχαριστώ. At the present moment... Αυτή τη στιγμή. Τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση Τις έχουμε χαρακτηρίσει και άλλωστε περιμένουμε ότι θα εφαρμοστούν 100% με τη μέγιστη αποφασιστικότητα. Τις χαρακτηρίσαμε λοιπόν ως και πιστικές και θαραλές. Επίσης, θεωρώ ότι, είναι υπόθεση βάσος αν θέλετε την οποία έχουμε αναπτύξει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι και οι φορείς της αγοράς και τα δημοσιονομικοί οργανισμοί, χρηματοπιστικοί οργανισμοί καλύτερα και ως, όλη η αγορά θα συμφωνήσει επίσης ότι είναι πιστικά αυτά τα μέτρα. Και γι' αυτό θεωρώ εγώ, μέσα στην υπόθεση αυτή που εργάζομαι, που επεξεργάζομαι καλύτερα, ότι δεν θα έχουμε δυσκολία τη στιγμή που θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα, τα έκτακτα μέτρα. Δεν θα έχουμε τέτοιου είδους δυσκολία διότι δεν θα υπάρχει η υποβάθμιση αυτή της υπογραφής της Ελλάδος. Εάν τυχόν και αποδειχθεί ότι αυτή η υπόθεση παρά ήταν αισιόδοξη, πράγμα το οποίο εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβεί, τότε θα εξετάσουμε την κατάσταση. Αλλά ε, σε αυτή τη χρονική στιγμή εγώ θεωρώ ότι βαδίζουμε προς αυτήν την εξέλιξη. Και πάλι με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται η αξιοπιστία του, του προγράμματος ανάκαμψης αναγνωρίζεται, πιστεύω, και θα αναγνωριστεί σταδιακά και από τις αγορές και από όλους τους παράγοντες. Ευχαριστώ. Ούντο Μπούλμαν. Πρόεδρε, έχω τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Μιλήσατε για, τις... για τα δάνεια στην Ευρωζώνη και βέβαια αναφέρεστε λίγο και στην κατάσταση στα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν ε, στρεβλώσεις, υπάρχουν στρεβλώσεις κερδοσκοπικές. Βλέπετε κάτι συγκεκριμένο εσείς στην υπόθεση αυτή την οποία περνάμε, κάποιους παράγοντες ή προϊόντα στρέβλωσης που δεν είναι αποδεκτά και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Και επίσης γίνεται μια συζήτηση περί ανάγκης ενδεχομένως εκδίωξης από την Ευρωζώνη ή μια ευρωζώνη αλλά κάρτα ενδεχομένω, από την οποία διώχνουμε όποιον ε, διαπράττει σφάλμα ή υποχρεούται να αποχωρήσει μέχρι ότου ε, μπορέσει να επανέλθει έχοντας διορθώσει τα εσφαλμένα. Ποια είναι η θέση η δική σας. Και τρίτη ερώτηση. Μιλήσατε για ανισορροπίες που βρίσκονται και μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλήσατε και για κράτη τα οποία έχουν μεγάλο ισοζύγιο εξαγωγών, πλεόνασμα εξαγωγών ή και μεγάλη παραγωγή και ερωτώ τι θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε μια σχετικά φρόνιμη οικονομική πολιτική στην δεδομένη οικονομική κατάσταση και πέραν βέβαια των όσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρώτη ερώτηση. Για τα σπρέντα, αν σας καταλαβαίνω σωστά, έτσι. Δεύτερο, η ερώτηση για το αν θα μείνει κανείς ή αν θα ιδιοκθεί κανείς από, το, από την Ευρωζώνη. Και τρίτη ερώτηση για τα πλεονάσματα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα λίγο πολύ. Για την πρώτη ερώτηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν διανοούμε να διατυπώσω ε, κατηγορίες έναντι αγορών ή μέσων. Ε, ή του CDS με βάση κάποιες συγκεκριμένες, της Επιτροπής Παρακολούθησης δηλαδή, ε, με βάση κάποιες συγκεκριμένες και στιγμιαίες παρατηρήσεις. Υπάρχουν δημοσιονομικοί φορείς, υπάρχουν ε, παράγοντες και οργανισμοί χρηματοπιστωτικοί και όχι μόνο τράπεζες πολύ πιο διαφανής. Υπάρχει ο ρόλος της ανάπτυξης των οικονομικών των χρηματοπιστωτικών μέσων και των παραγόγων κατά τρόπο πιο, πιο διαφανή. Αυτό είναι το καθήκον μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, προχωρούμε με αποφασιστικότητα, έχουμε πολλή δουλειά και πιστεύουμε ότι ακόμα πολλά μένουν να γίνουν. Αλλά δεν πρέπει και να μπερδευόμαστε και να συγχαίουμε όλα αυτά με την ε, γενικότερη εικόνα της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι όλοι οι φορείς είναι σε θέση να αναγνωρίσουν το τι κάνει, το τι πράττει η Ελλάδα και τότε θα μειωθεί και το spread, το περιθώριο δηλαδή, κατά ουσιαστικό τρόπο. Αυτό επίσης θεωρώ εγώ ότι θα συμβεί. Αυτή είναι η υπόθεση εργασίας με την οποία εργάζομαι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω πάρει τα πράγματα ελαφρά. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, οπωσδήποτε. Το να παραμείνει κανείς μέσα ή έξω από τη ζώνη ευρώ. Η ζώνη του ευρώ δεν είναι à la carte. Μπαίνει ένα κράτος με στη ζώνη ευρώ για να έχει μια κοινότητα πεπρωμένου. Μοιράζεται τη μοίρα του με τους άλλους με, αυτή την επιλογή ερχόμαστε και μπαίνουμε μέσα, με αυτή την επιλογή αναπτύσσουμε και αναπτύξαμε και τις συνενέσεις μέσα στη ζώνη του ευρώ. Έχουμε μια κοινότητα πεπρωμένου και στα γερμανικά σας το λέω και στα γαλλικά σας το λέω και στα αγγλικά σας το λέω. Σας είπα ότι θεωρώ παράλογη την υπόθεση του να εγκαταλείψει κανείς τη ζώνη του ευρώ. Άλλωστε νομικά δεν επιτρέπεται. Άρα δεν τίθεται το ερώτημα σήμερα, είναι non-question. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι ζήτημα για αύριο, διότι θεωρώ ότι δεν ευθυγραμμίζεται με την ουσία την ίδια, με την πεμπτουσία της ζώνης του ευρώ. Και αν κάτι πρέπει να ενισχύσουμε, είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση της ευθύνης. Η ευθύνη την οποία καλείται κανείς να επιτελέσει και έναντι των εταίρων του όταν ο εταίρος του δεν συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Με τον έλεγχο δηλαδή των εταίρων των ομοτήμων. Επίσης, χώρες που έχουν μια σχετικά καλή ανταγωνιστικότητα. Επειδή είναι καλή ανταγωνιστικότητά τους, έχουν ένα ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών πλεονασματικό. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να τις επικρίνουμε. τρεις ή τέσσερις χώρες. Αν κοιτάξουμε τι έχουν προσφέρει στην Ευρωζώνη, αυτές που έχουν τα πλεονασματικά ίσως για τα τελευταία 10-11 χρόνια. Τι έχουν προσφέρει λοιπόν ζώνη του ευρώ. Έχουν γενικό ε, πληθωρισμό κάτω του μέσου όρου. 1,95% πληθωρισμό προβλέπουμε για τα πρώτα 12 χρόνια του ευρώ. Ακριβώς αυτό το οποίο είχαμε προσδιορίσει ως σταθερότητα των τιμών. Πολύ κοντά στο 2. Κάτω από το 2, πολύ κοντά στο 2. Άρα θα έχουμε επιτύχει αυτή τη σταθερότητα των τιμών. Ναι. Τώρα, εάν κάποιες χώρες είχαν υψηλότερο πληθωρισμό, η νομισματική μας πολιτική θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή. Άρα, πρέπει να αναγνωρίσουν αυτό το δεδομένο όλες οι χώρες. Θα είχαμε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, αν ορισμένες εκ των χωρών του ευρώ δεν είχαν συμπεριφερθεί Όπω συμπεριφέρθηκαν. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά και άλλε χώρε μέλη. Και αυτό ισχύει και για το ισοζύγιο ε, τρεχόντων λογαριασμών. Ερωτώ λοιπόν, για το τρέχον ισοζύγιο δηλαδή, πώς θα είχαμε χρηματοδοτήσει το, το έλλειμμα του ισοζυγίου άλλων κρατών, αν δεν είχαν εκείνοι ισοσκελισμένο τον προπολογισμό τους. Έτσι μόνο μπορούσαμε να βοηθήσουμε εκείνους που είχαν πρόβλημα. Μπορέσαμε χάρη σε αυτούς, γιατί κάποιοι δεν συνέβαλαν στις ανισορροπίες. Έχοντας πλεόνασμα, χρηματοδότησαν το έλλειμμα των άλλων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι ικανοποιημένο από αυτό το καθεστώς και ότι θα ήθελα να είναι μόνιμο, θα πρέπει όλοι λίγο πολύ να κινούμαστε κάπου στο μέσον όρο, μακροπρόθεσμα και μακροχρόνια, και γι' αυτό απευθύνω και έκκληση, έτσι ώστε οι όχι πολύ καλά λειτουργούσες οικονομίες, εκείνε που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να έχουν καλύτερο ισοζύγιο, να είναι πιο ισοσκελισμένε και ω εκ τούτου και πιο ανταγωνιστικές και προσμένω ότι αυτοί που θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα δεν θα είναι πάντα οι καλύτεροι από τους άλλου, γιατί μακροπρόθεσμα δεν θα έχουν αρκετό χώρο μέσα στο περιορισμένο χώρο του ευρώ. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως και τον πληθωρισμό, εμείς για τα πρώτα 12 χρόνια της ύπαρξης του ευρώ, επαναλαμβάνω, εάν μέχρι τα τέλη του έτους δεν διαψευστούν οι προβλέψεις μας, το 1,95% που προβλέπουμε, που είναι λίγο καλύτερο από ό,τι είχε παραδείγματι για την ίδια προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη 12 ετία η Bundesbank της Γερμανίας ή και την προηγούμενη 20 ετία αν θέλετε. Άρα είμαστε αρκετά ευθυγραμμισμένοι πιστεύω με ένα κατάλληλο, με ένα σωστό επίπεδο ε, σταθερότητα τιμών. Αυτό που παγκοσμίω γίνεται αποδεκτό στο το βέλτιστο επίπεδο σταθερότητα τιμών. Πολύ σύντομα λέει ο κ. Μπούλμαν. Δηλαδή, απάντηση στην ερώτησή μου είναι ότι καλείται και τα άλλα κράτη-μέλη να αναπτύξουν πλεονάσματα. Απάντηση όχι. Θα έλεγα ότι μακροπρόθεσμα όλες οι χώρες, όλες οι οικονομίες, αλλά προσοχή έτσι, γιατί θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη δημογραφική κατάσταση κάθε χώρας, χώρα η οποία έχει κακή δημογραφική εξέλιξη, ασφαλώς θα έχει πλεόνασμα κάποιου συγκεκριμένου όγκου, ενώ μια χώρα η οποία έχει μια πολύ δυναμική δημογραφική εξέλιξη θα έχει τελείω διαφορετική εικόνα να παρουσιάσει. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Έτσι. Άρα τηρουμένων των αναλογιών θα πρέπει όλε οι χώρε λίγο πολύ να ε, κυμαίνονται στον μέσο όρο του πληθωρισμού της, ζώνη ζώνης του ευρώ. Και πάλι όπως είπα λαμβανωμένη υπόψη και των δημογραφικών στοιχείων. Μεγαλύτερο ή μικρότερο πλεόνασμα θα πρέπει να παρουσιάζουν ανάλογα με τις δημογραφικές τους συνθήκες, αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, θα πρέπει ε, αυτό να καταλήγει σε ένα γενικό ισοζύγιο, ισοσκελισμένο μάλλον, μια γενικά ισοσκελισμένη εικόνα για τη ζώνη του ευρώ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωραία. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, ο χρόνος περνάει όμως. Παρακαλώ. Κύριε Τρισέ, εδώ είμαι. Λέει ο κύριος ε, Σκλούνα. Θυμάμαι πως ε, επιμένατε υπέρ του συμφώνου σταθερότητα, όταν κάποιε χώρε θέλανε να αποδυναμωστεί, αλλά οι υπουργοί κάποια στιγμή αποφάσισαν να μην δεχτούν την πρόταση της Επιτροπής να μην γίνεται έλεγχος στι στατιστικέ των δημοσιονομικών. Εσείς τώρα είσαστε ευτυχεί, δηλαδή αν δείτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκεί έχουν πιο ευρύτερο πεδίο Ωραία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μιλάει με τις κεντρικές τράπεζες, η Κομισιόν μιλάει με υπουργού, Γιατί όμως να μην ανοίξουμε κάπως και με άλλους παράγοντες, με την αντιπολίτευση, με τα συνδικάτα, με ειδικού, ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία και δεδομένα. Τέλος, είστε ευτυχείς με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα πλαίσια της διαδικασίας αντιμετώπισης του λίματος. Τρισέ. Ε. Πρώτα απ' όλα, όταν αποφασίστηκε να μην γενικευθεί ο έλεγχος, δεν ήμασταν ευχαριστημένοι. Η έλεγχη επιτόπου, ε. Και προσδοκώ να ληφθεί η σωστή απόφαση σήμερα. Είναι αναγκαίο. Πλήρης διαφάνεια χρειάζεται. Και πλήρης κατάργηση των παιχνιδιών που παίζονταν στο παρελθόν. Είναι ζωτική σημασία Ξεκάθαρο. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Έχουμε επιμονή μου βάσεως διάλογο εμείς με οικονομολόγους. Συμμετέχουμε δραστήρια και σε συνέδρια, σε συζητήσεις που γίνονται εκεί και στην έδρα μας έρχονται, οπότε είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο συμμετέχουμε και στον μακροοικονομικό διάλογο με συνδικάτα στην Ευρώπη, τακτικά. Και έτσι, από αυτή την άποψη, το κάνουμε. Βέβαια, είμαστε ανεξάρτητοι. Και εφόσον είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον κόσμο εμείς. Και λογοδοτούμε στην κοινή γνώμη. Οπότε δεν βλέπω γιατί να μην έχουμε τέτοιο διάλογο, να μην πηγαίνουμε, να απαντάμε στις ερωτήσεις που μας ρωτάει ο κόσμος. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, εμείς το θέλουμε. Απάντηση, έτσι δεν είναι. Για το υπερβολικό έλλειμμα, τη διαδικασία όσον αφορά το υπερβολικό έλλειμμα, αν είσαστε ικανοποιημένο ή όχι, ε, υπενθυμίζει η πρόεδρο στον κύριο Τρισέ την ερώτηση. Τρισέ, πρέπει να ενισχύσουμε την εφαρμογή της διαδικασίας όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εννοείται ότι είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει όμως να είμαστε υπερβολικά αρνητικοί, επιτρέψτε μου όσον αφορά την Ευρωζώνη, διότι βλέπετε υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη που αποτελεί βέβαια ένα περίπλοκο σύστημα οργάνων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο κλπ. Έχουμε λοιπόν την τάση μερικές φορές να επικεντρωνόμαστε υπερβολικά σε πράγματα τα οποία δεν πάνε καλά και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα και θα έπρεπε να λειτουργούν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά όμως δείτε την Ευρωζώνη σαν μια παγιωμένη οικονομία. Όπως όταν είπα ότι υπάρχει ισορροπία σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είμαστε εμείς που ενισχύουμε τις ανισορροπίες παγκοσμίω, όχι. Λοιπόν, αν δείτε τα δημοσιονομικά της Ευρώπης, το έλλειμμα είναι 7% του ΕΠ στην Ευρωζώνη. 7% του ΕΠ. Βέβαια, δυστυχώς, ορισμένοι έχουν το διπλό. Ορισμένοι είναι κάτω από αυτό. Πάντως, ο μέσος όρος είναι 7%. Ποιο είναι το επίπεδο το αντίστοιχο στις ΗΠΑ. 10,5%. Άρα 3,5% παραπάνω από το δικό μας το έλλειμμα της Ευρωζώνης. Η Ιαπωνία 10,5% κι αυτή. Πάλι 3,5% παραπάνω από το έλλειμμα της Ευρωζώνης. Οι δύο άλλοι μεγάλοι στην οικονομία παγκοσμίω, έτσι. Και θα μπορούσα να πάρω και άλλα παραδείγματα και να βρω και άλλους παραπάνω από το δικό μας το επίπεδο στην Ευρωζώνη. Και αυτό το λέω για να σημειώσω ότι ακόμα κι αν δεν εφαρμόζεται αρκετά καλά και λιγότερο καλά ε, σε ορισμένες χώρες. Είναι προφανές αυτό. Παρ' όλα αυτά, στο σύνολο το σύμφωνο σταθερότητας έπαιξε κάποιο ρόλο και μας βοήθησε να μην βρισκόμαστε στα επίπεδα που έχει έλλειμμα η Αμερική και η Ιαπωνία σήμερα. Σιλβί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σε πολλές γλώσσες αναφέρατε το κοινή μοίρα. Δεν νομίζω ότι ο ευρωπαϊκός τύπος όμως λέει τα ίδια. Διότι θεωρώ ότι πολλοί ξεχάσανε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα από κοινού. Εγώ έχω τώρα μία φιλοσοφικού χαρακτήρα ερώτηση. Μας λέτε έχουμε μία κοινή μοίρα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε κανόνες και λίγο peer pressure για να προχωρήσουν όλα αυτά. Ε, είναι δύσκολο να... Δύσκολα δόθηκαν ε, δόθηκε ο δωδεκάλογος στο συνάστον ε, στο Μωυσή. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ε, ότι παρά τον δωδεκάλογο ενώ συνεχίζει ο κόσμος να αμαρτάνει ότι έχοντας εμείς αυτή την peer pressure θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι και θα συνεχίσουμε να συνεχίζουμε την πολιτική για το ευρώ η οποία δεν θα βλαφθεί για το μέλλον. Η πίεση των ομοίων, ε, από, ε, pression de από τα παλιά, από τα αρχαία αγγλονορμανδικά θα πρέπει να προέρχεται αυτό ή από τα αρχαία αγγλικά. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να μεταδώσω εδώ από την Κεντρική Τράπεζα είναι ότι σημεριζόμεθα πολύ περισσότερο ένα κοινό, μια κοινή μοίρα, πολύ περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι φανταζόμασταν ότι συμμεριζόμασταν. Και η κρίση αυτή είναι η χειρότερη κρίση μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ίσως και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ζούμε αυτό και αν δεν υπήρχαν οι πολύ θαραλέες αποφάσεις ε, των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων ε, αυτή η κρίση ε, δεν δε θα είχαμε βγει από αυτή την κρίση και αυτή η κρίση είναι, βγάζει στην επιφάνεια πράγματα και γυρνάμε στις ε, πηγές γυρνάμε στους πατέρες ιδρυτές του ευρώ ότι μοιραζόμαστε μια κοινή μοίρα και οι 27 την κοινή μοίρα θέλουν να μοιραστούν. Κοινή μοίρα δηλαδή ευημερία και ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και την επιτυχία. Και η επιτυχία δηλαδή ήταν πραγματικά λαμπρή και το λέω εδώ υπό το όμα των εκλεγμένων εκπροσώπων του ευρωπαϊκού λαού που τα ελέγχουν όλα αυτά. Αυτό το οποίο λοιπόν έχουμε σήμερα από φιλοσοφικής πλευράς που είναι η απόλυτη κατανόηση του τι ζούμε, του τι βιώνουμε. Τώρα, μία χώρα που είναι το 2,5% του ακαθαρίστου προϊόντος της Ένωσης, δηλαδή ένα πυρελάχιστο τμήμα της Ένωσης. Και το πρόβλημά του γίνεται κατανοητό το και το νιώθουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης και έχει επιπτώσεις και στις, ε, στις άλλες κράτη-μέλη δείχνει ότι έχουμε αυτή την κοινή μοίρα, αυτή τη συλλογική μοίρα που είναι ουσιαστική. Το μήνυμά μας λοιπόν είναι ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, συνολικά τις ευθύνες του, σε κάθε περίοδο, όποια περίοδος και να είναι. και θα έλεγα να ασκήσει και την φιλική πίεση προς τις κυβερνήσεις που είναι πιο σθεναρές, πιο αμετάκλητες, σκεπτόμενοι το κοινό καλό, όπως το πρόβλεψαν οι συνθήκες, όπως το πρόβλεψαν οι πατέρες ιδρυτές και που θεωρούμε και εμείς ότι πρέπει να το κάνουμε. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και εμεί είμαστε εντελώ ομοσπονδιακό θεσμικό όργανο, έχουμε ένα νόμισμα και θέλουμε να προασπιστούμε την αξιοπιστία ενός νομίσματος έναντι των 330 εκατομμυρίων Ευρωπαίων συμπολιτών. Okay. Η σχέση μεταξύ νομισματική και δημοσιονομική πολιτικής ε, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εξέλιξη ευρωπαϊκής οικονομίας και ω εκ τούτου και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν λοιπόν θέλει να παραμείνουν τα ποσοστά του πληθωρισμού κοντά και κάτω από το 2% για το μέλλον, τι θα πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσει σε σχέση με την με τους ε, κινδύνους, ε, ο δανεισμός τους να οδηγήσει σε πιέσεις ε, στον πληθωρισμό από τις αγορές. Επομένως, τι είδου δημοσιονομική πολιτική πιστεύετε ότι θα χρειαστεί. Και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να συντονίζει, να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή αυτών των δανείων των κρατών μελών και ενδεχομένως να έχει και ένα ρόλο προγραμματισμού των προθεσμιών αποπληρωμής. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, όπως γνωρίζετε, το ΕΚΟΦΗΝ επί τη βάση της εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επί τη βάση της αποδοχής από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, της έγκρισης μάλλον των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, τους έχει λάβει μια σειρά αποφάσεων. Και εδώ, όπως είπα και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, αυτό που ζητούμε είναι πλήρης τήρηση των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί. Και από ό,τι θυμάμαι εγώ, η νέα συνθήκη ορίζει ότι οι εταίροι, οι ομότιμοι, οι ομόλογοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και η εν λόγω χώρα δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Αυτά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ορίζει η νέα συνθήκη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε λογικοί έτσι ώστε να μην παραφορτώνουμε την νομισματική μας πολιτική, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξουμε και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη. Γιατί η εμπιστοσύνη, το αίσθημα της εμπιστοσύνης έχει τεράστια σημασία σε αυτή τη χρονική στιγμή. Είναι απολύτως απαραίτητο να πείσουμε τους πολίτες, τα νοικοκυριά, τους επιχειρηματίες, τους οικονομικούς παράγοντες εν γέννη, ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον των ίδιων τους των επιχειρήσεων και στο μέλλον των ίδιων τους των οικοκυριών. Ότι δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε παραφορτώσει με τεράστια χρέη, με αφόρητες ε, ε απαιτήσει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία πιστεύω και κυρίως για τις χώρες οι οποίες έχουν το άμεσο και συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά ισχύει για τους πάντες. Όχι μόνο βέβαια για τη ζώνη του ευρώ, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ούτε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο, αλλά για όλες τις χώρες του βιομηχανικού κόσμου, του εκβιομηχανιστέντο κόσμου. Αυτό είναι όλο. Εγώ θα έλεγα επίσης να μην ε, παρεμβαίνει υπερβολικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως προς το ε, υποστήριξη, το αρρωγή στο συντονισμό σε τέτοιου είδους ε, προγράμματα ή τον τρόπο με τον οποίο θα, χειρίζεται ένα κράτος το, τα δάνειά του ή τη νέα του δανειοληπτική δραστηριότητα. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι με ξαφνιάζει το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες χώρες επειδή ε, βρήκαν ελκυστικά τα βραχυπρόθεσμα ε, επιτόκια είχαν την τάση να μειώσουν τη διάρκεια των χρονίων τους ε, δανείων, πράγμα το οποίο βέβαια είναι λάθος γιατί οδηγεί σε πιο μεγάλη ε, αστάθεια ή ενδεχομένως καθιστά την οικονομία της χώρας πιο ευάλωτη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται μια χώρα, μια κυβέρνηση, το υφιστάμενο της χρέο, τα δάνεια που έχει αναλάβει. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν είναι δουλειά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή εσδήποτε κεντρική τράπεζα, αν μου επιτρέπετε, να δεσμεύεται, να, παρεμβαίνει μάλλον στον χειρισμό τέτοιου είδου οικονομικών συνθήκων. Ο κύριος Χουντής, παρακαλώ. Um, Ζητώ συγγνώμη. Λυσμόνισα τον Πασκάλ. Με συγχωρείτε κύριε Χουντή, Λυσμόνισα ότι είχα ε, προηγουμένως ε, σημειώσει τον Πασκάλ πριν από σας. Ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα κύριε Τρίσε, είμαι. Λοιπόν, να σταθώ λίγο στην ερώτηση του κυρίου Μπούλμαν σχετικά με τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα του ισοζυγίου. Ήταν ενδιαφέρουσα η απάντηση και βρίσκεται και στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαχείρισης. Άμα κανείς δει πως εξελίσσονται τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα στη ζώνη ευρώ, βλέπουμε αύξηση των ελλημάτων από τη μια και των πλεασμάτων από την άλλη. Επειδή μιλήσαμε πολύ για νούμερα, ξέρετε ότι 14% του ΑΕΠ είναι το έλλειμμα του ισοζυγίου της Ελλάδας, είναι πραγματικά ασήκωτο και από την άλλη έχετε ένα πολύ ψηλό πλεόνασμα της Γερμανίας που είναι 7% του ΑΕΠ. Λοιπόν, μπορείτε εσείς ε, ως ε, πιλότος ε, των οικονομικών δεν μπορείτε να έχετε μία ενιαία νομισματική πολιτική όταν έχουμε τέτοιου είδους διαφορές κάθε χρόνο που θα εντείνονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, και η οι Γερμανοί, δεν έχουν ανατίμηση του Μάρκου γιατί δεν υπάρχει πλέον το Μάρκο και οι Έλληνες δεν μπορούν να υποτιμήσουν τη δραχμή τους γιατί δεν έχουν πλέον δικό τους νόμισμα. Λοιπόν, ρωτώ, εσείς ε, τι φαντάζεστε ως ε, μέσο χωρίς να έχουμε καμία ηθική ε, εκφορά απόψεων, τι φαντάζεστε ως μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κρατιέται η ισορροπία μέσα στη ζώνη ευρώ. Για να μην έχουμε αυτές τις ανισορροπίες που αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη του ευρώ. Λέτε ε, που να μην αμφισβητούν ε, το λόγο ύπαρξης του ευρώ. Αυτή είναι η πρόταση που δεν προσυπογράφω διότι υπάρχουν μηχανισμοί σε αυτήν την ε, τεράστια υπηρετική ζώνη ενιαίου νομίσματος, υπάρχουν διορθωτικοί μηχανισμοί μέσα από το κανάλι ανταγωνιστικότητας το οποίο λειτουργεί και το οποίο όμως μπορεί να λειτουργήσει πολύ αργά ε, και σε αυτό συμφωνώ ότι στο μεταξύ μέχρι να λειτουργήσει διαφορές είναι μεγάλες. Έχουμε τις επαφές μας όμως με την Ευρωομάδα και από το 2005 εγώ υποδεικνύω στα μέλη της Ευρωμάδας ότι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να περιφρουρήσουν είναι η, σχετική, εξέλιξη της σχετικής ανταγωνιστικότητας, δηλαδή ε, κόστος ε, μονάδα, μονάδα παραγωγής ε, κλπ. Δηλαδή, εμείς τα 10 χρόνια του ευρώ προσπαθήσαμε να ανασύρουμε διδάγματα για το μέλλον και τότε εγώ είχα επιμείνει ότι πέρα από την προσεκτική παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών θα πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά και την σχετική ανταγωνιστικότητα και την τις επιπτώσεις που έχει αυτή η σχετική ανταγωνιστικότητα στο τρέχον ισοζύγιο για τα πλεονάσματα και, το, ε, και τα ελλείμματα. Και μία χώρα με τόσο χαμηλή δημογραφική ανάπτυξη όπως η Γερμανία να έχει τόσα πλεονάσματα, η δημογραφική ανάπτυξη και αυτή παίζει ρόλο. διότι εκεί λειτουργεί το, το σύστημα λέγοντας ορίστε θα βάλουμε στην άκρη για να διαφυλάξουμε το σύστημα των συντάξεων κλπ. Αυτό ισχύει ε, για πολλούς από τις, πολλές από τις χώρες της Ευρωζώνης. Για να επανέλθουμε στην καρδιά του ζητήματος είναι το θέμα της ε, σχετικής ανταγωνιστικότητας και θα μιλ, πω τα ίδια πράγματα όπως έλεγα πριν για το μόνιμο καθεστώς. Όταν έχουμε εμείς αυτό το σταθερό καθεστώς στη ζώνη ευρώ έχουμε μια, έναν πληθωρισμό μεταξύ του 1 ή του 2%. Και εκεί έχουμε ε, σταθερότητα των τιμών, έχουμε ένα παγκόσμιο benchmark, ε, ε, market, έχουμε Έχουμε 2% τα ίδια θα έλεγε και ο Αμερικάνος συνάδελφος άμα του λέγατε ας πούμε ποια είναι μια άνετη ζώνη πληθωρισμού θα σας έλεγε λιγότερο από το 2% θα έλεγε ίσως δεν θα έλεγε ε, σίγουρα εμείς λοιπόν εγγυόμαστε αυτό το πράγμα οι εθνικοί πληθωρισμοί θα πρέπει να κυμαίνονται γύρω από αυτόν το μέσο όρο αν οι εθνικοί πληθωρισμοί είναι πάντα υψηλότεροι, σίγουρα υπάρχει απώλεια ανταγωνιστικότητας χρονιά με τη χρονιά. Δεσμεύω λοιπόν όλες τις εθνικές κυβερνήσεις και σίγουρα αυτές οι οποίες βρίσκονται σε μια κατάσταση με, με, με, μέσης ανταγωνιστικότητας να τα διορθώσουν όλα αυτά. Είτε να είναι σε επίπεδο δηλαδή του δικού της δικής μας σταθερότητας τιμών και αυτό έκανε και η Γερμανία. Η Γερμανία μπήκε στο ευρώ σε μια κατάσταση μη σχετικής ανταγωνιστικότητας μετά από την επανένωση. Είχε προβλήματα ανταγωνιστικότητας για πολλά χρόνια και είχε εθνικό πληθωρισμό λίγο χαμηλότερο από ό,τι αυτόν τη ζώνης. Ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό δεν είναι ανορμάλ. Είναι η κανονική λειτουργία ενός, ε, μιας μεγάλης υπηρετικής ζώνης με νέο νόμισμα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί, ε, να βελτιώνεται και να παρακολουθείτε η σχετική ανταγωνιστικότητα. Εσείς το γερμανικό πλεόνασμα μην το βλέπετε ως υπερανταγωνιστικότητα. Η Γερμανία πρέπει να προετοιμάσει το δημογραφικό της μέλλον. Ίσως πρέπει να ακούσουμε κι άλλες ερωτήσεις. Κύριε Χούντι, τώρα εσείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή όπως παραδεχτήκατε και όπως διαπιστώσαμε όλοι είναι η περίοδος που ακούμε πολλά και αντιφατικά πράγματα. Θέλω να κάνω τον εξής συλλογισμό. Μέχρι πρόσφατα και εσείς όταν ξέσπασε η κρίση λέγατε ότι κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνη της. Προσφάτως μεταξύ άλλων και εσείς αν δεν κάνω λάθος μιλάτε ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος μηχανισμός στήριξης, υποστήριξης και ούτω καθεξής. Σας ερωτώ, αυτή η προσπάθεια για στήριξη που είναι έξω από τις συνθήκες στη βάση ποιας θεσμικής, θεσμικού πλαισίου θα γίνει και με ποιους όρους. Και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα παρατείνει την εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Έχει δώσει 11 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρουμε αν έχουν πάει στην πραγματική οικονομία, μένουν άλλα 16. Σας ερωτώ, ποια είναι η γνώμη σας να συνεχίσει να δίνει, να ενισχύει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών η ελληνική κυβέρνηση τη στιγμή που κάνει αγώνα το κεντρικό πρόβλημα να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα. Θα συμβουλεύατε δηλαδή τον Υπουργό ε, Οικονομικών να συνέχισε μια τέτοια ενίσχυση των τραπεζών τη στιγμή που έχει αυτές τις δυσκολίες. Uh, Ήδη έχω πει ότι Πριν δεν το Για, τις, ε, για την περιοχή της Ευρωζώνης μίλησα πριν για ένα δάνειο χωρίς ειδικού όρους εφόσον υπάρχουν οι όροι και Αν δεν είναι μερικού το μέσο αυτό. Εάν αντιστοιχεί σε άμεση απειλή για την ελόγω χώρα και αν και εφόσον έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. όπως είπε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα θυμόσαστε ότι είπε ότι οι χώρες της Ευρωζώνης θα πάρουν συντονισμένες δράσεις εφόσον χρειαστεί για τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη, γιατί υπάρχει απειλή στην Ευρωζώνη στο σύνολό της. Αυτό το είπαμε λοιπόν και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Όσον αφορά τώρα το θέμα της στήριξης που αποφασίστηκε από τις διάφορες κυβερνήσεις για τη δικιά τους δημοσιονομική σφαίρα, πράγματι υπήρξε μεγάλη στήριξη. Ξέρετε ότι η Κεντρική Τράπεζα κοίταξε τη στήριξη για, την τράπεζες, για τις τράπεζες, φτάσαμε στο 25% του ΑΕΠ, όχι μόνο για τις τράπεζες και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένε Πολιτείε το ίδιο. Μιλάμε για την ίδια τάξη μεγέθους. Η στήριξη αυτή που αποφασίστηκε από τις κυβερνήσεις και που είναι επιπλέον από αυτά που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί απαραίτητα και ούτε σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και κέρδο σε πολλές περιπτώσεις. Όμως ήταν αναγκαίο να κινητοποιηθεί αυτό το επίπεδο. Όντως, σε μικρές χώρες υπήρξε μια αντιστοιχία με την στήριξη που δόθηκε σε επίπεδο και άλλων βιομηχανικών χωρών, ΗΠΑ κλπ. Η κυρία Τζαβέλα. Κύριε Πρόεδρε, οι ελληνικές τράπεζες είναι ουσιαστικά υποκαταστήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην παρούσα περίοδο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό και υγιέστατο. Δόξα τω Θεώ οι τράπεζες στην παρούσα περίοδο οι ελληνικές δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Προληπτικά τώρα τοποθετούμε κύριε Πρόεδρε και το τονίζω προληπτικά. Όσο παρατείνεται η εκκρεμότητα με την κρίση στην Ελλάδα, εκφράζω την ανησυχία μήπως οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάσουν πιθανό πρόβλημα ρευστότητας. Εφόσον λοιπόν οι τράπεζες αυτές είναι ουσιαστικά υποκαταστήματα της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, θα δηλώνατε ότι σε περίπτωση που παρουσιάσουν ρευστότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσιάσουν πρόβλημα ρευστότητας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες. we will of course apply all our rules as uh, we... Βεβαίως θα εφαρμόσουμε όλους τους κανόνες όπως πράξαμε και με την Ιρλανδία και με όλες τις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ. Είναι αυτονόητο αυτό, δεν χρειάζεται να το πούμε. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Γκέρι, πρόεδρε, με μεγάλη χαρά σας βλέπουμε και πάλι εδώ. Κύριε Τρισέ, όπως ίσως έχετε υπόψη, έχουμε στο πρόγραμμά μας τη συζήτηση για το σύστημα εποπτείας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι έχετε να πείτε για το ε, Συμβούλιο Διαχείρισης Συστημικών Κινδύνων που θα υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για συμφωνώ σε αυτό. Αλλά πείτε μου παρακαλώ για τα μέσα που θα έχει σε θέση του αυτό το Συμβούλιο. Πώς θα μπορεί δηλαδή να κάνει μια καλή δουλειά και να μας προειδοποιεί εγκαίρως για τους κινδύνους, τους επερχόμενους κινδύνους. Πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό το συμβολιό; Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη. Πάλι για το ίδιο συμβολιό; Οι τροπολογίες που έχουμε εμείς καταθέσει σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έλεγε ότι θα υπάρχουν πέντε ε, που θα προσδιορίζονται από μια διευθυντική επιτροπή του, Γενικού, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, χωρίς όμως να ορίζονται αναλογίες συγκεκριμένε και έτσι υπάρχει μια ουγγροπολωνική τροπολογία στη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία ζητεί να υπάρχει εκπροσώπηση κατά αναλογία μελών ευρωζώνης και εκτός ευρωζώνης. Νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η τροπολογία, γιατί η κρίση μας επηρεάζει όλους και όχι μόνο τα μέρη της ευρωζώνης. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και εκπρόσωποι πραγματογνωμόνες από τα κράτη που βρίσκονται έξω από τη ζώνη του ευρώ. Και γι' αυτό δεν ήθελα να μου πείτε αν υποστηρίζετε και σε αυτήν την ιδέα. Κύριο Στρισέ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, το Συμβούλιο αυτό συστημικών κινδύνων θα έχει βέβαια ως κύριο μέσο στη διάθεσή του την δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις 27 κεντρικές τράπεζες, εθνικές κεντρικές τράπεζες, που θα έχουν και βέβαια τους διοικητές τους, αλλά και την ε, υλικοτεχνική τους υποδομή στη θέση του Συμβουλίου και επίσης στα, στο δυναμικό του θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει το προσωπικό του από τα 27 κράτη-μέλη. Και με την παρουσία των αρχών των επικεφάλειες των διαφόρων αρχών, εν πάση περιπτώσει, με τη μικροεποπτεία και λαμβανωμένη υπόψη ότι θα έχουμε, λαμβανωμένη υπόψη ότι έχουμε παρόντες και τους διευθυντές, τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών και όλα αυτά και όπως άλλωστε προτάθηκε από τον Λαγοζιέρ και έγινε και δεκτό στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα βλέπουμε να το εξετάζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ε, συνεργασία από ό,τι βλέπουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς, πιστεύω ότι θα δοθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος έτσι ώστε να ε, διαμορφωθούν οι εργασίες αυτού του Συμβουλίου ε, Συστημικών Κινδύνων κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, γιατί αυτό χρειάζεται. Να μπορούμε να προβλέψουμε τους συστημικούς κινδύνους του μεγέθου που ανέφερα νωρίτερα. Για τι τροπολογίε στι οποίε αναφερθήκατε θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα νομικά πιθανό πρόβλημα, αλλά και πάλι δεν μπορώ εγώ να, να ε, τοποθετηθώ στις εσωτερικές συζητήσεις σας, έτσι, γιατί το κοινοβούλιο συζητεί αυτή την τροπολογία πλέον, όχι εγώ. Αλλά ε, αυτό που θα έβλεπα εγώ σαν πρόβλημα θα ήταν ότι η ζώνη του ευρώ ε, μεγενθύνεται σύντο χρόνο. Ξεκινήσαμε 11, έχουμε φτάσει να είμαστε 16 τώρα. αν αρχίσουμε να λέμε τρεις έξω, δύο μέσα, κινδυνεύουμε να χάσουμε την, ε, το συσχετισμό, να χάσουμε τον έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δύο χώρες που έχουν το opting out, το έχουν τον, τον αυτοαποκλεισμό από τη ζώνη του ευρώ. Επομένως θα πρέπει να σεβαστούμε τις δομές των 27, αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Φυσικά θα πρέπει να εκπροσωπεί τις δομές των 27 το Συμβούλιο αυτό. Εάν αυτό εννοείται με την τροπολογία, ασφαλώς και έχετε δίκιο. Απλώς δεν θεωρώ ότι είναι δεδομένο πως θα πρέπει να καταγραφεί μέσα στο νομικό αυτοκείμενο. Γιατί ίσως να μην βρίσκει τη θέση του και στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη όμως του ευρώ. Ο κύριος Κάρας. Mm. Πρόεδρε. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Είδαμε τον ε, Πρωθυπουργό της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Κρίσεως εδώ, και μας είπε ότι εάν ε, η Ελλάδα χρειαστεί να ακολουθήσει τους κανόνες ε, του Διεθνούς Οσματικού Ταμείου, δεν θα λάβει χρήματα. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα του Διεθνούς Οσματικού Ταμείου, δηλαδή η προσφυγή σε αυτό ώστε μακροπρόθεσμα να εξασφαλιστούν τα κονδύλια και ταυτόχρονα η ανάγκη να καλυφθεί το μέχρι τότε διάστημα. Εσεί τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και επίση είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα ότι δεν θέλει και δεν ζητάει χρήματα. Δύο μέτρα χρειάζεται και ζητάει. Την προστασία από τι παγκόσμιε χρηματοπιστωτικέ αγορέ και την κερδοσκοπία του, δηλαδή τα πολύ ψηλά επιτόκια στο δανεισμό που προσφέρεται στην Ελλάδα και ρωτώ τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ελλάδα και επιπλέον ερώτηση μιλήσατε για την, ε, για την Οικονομική Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν αρκεί για μια Οικονομική Ένωση. Τι χρειάζεται λοιπόν επιπλέον για να εξασφαλίσουμε μια Οικονομική Ένωση. Και σε σχέση με τα όσα είπε ο Επίτροπος Ρεν για την δημοσιονομική πολιτική τις τελευταίες ημέρες, τι έχετε να πείτε. Uh, Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι άμεσο. Είναι το πρόγραμμα ανάκαμψης της Ελλάδας και εφαρμογή του. Είναι θέμα της αξιοπιστίας που πρέπει να ανακτήσει η Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα που επήγει. Τώρα μία νέα δομή. Φυσικά και είναι κάτι που πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα. Αν κατάλαβα καλά αυτό που λέτε, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε, γενικά το νομισματικό δεν μας αρέσει πολύ σαν όρος. Ένα νομισματικό Ινστιτούτο στην Ευρώπη τώρα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε τι θα κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Θα οργανώνει ακριβώς αυτήν την ε, περίπτωση δικής στήριξης. Για να ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι όροι του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Οι προϋποθέσεις που ανέφερα για να δίνεται αυτού του είδους ειδική βοήθεια στην Ελλάδα σήμερα θα είναι ακριβώς ίδια και στο μέλλον. Πάντως είναι η πρόταση που έγινε από μια κυβέρνηση που πρέπει να μελετηθεί. Η συγκεκριμένη δηλαδή πρόταση να μελετηθεί και από τους υπόλοιπους. Το μόνο σημείο για το οποίο θα ήμουν αρνητικός, όπως θα το έχετε ήδη καταλάβει, είναι η ιδέα του να βγει μια χώρα, να διωχτεί μια χώρα. Δεν πιστεύω ότι ταιριάζει με την ίδια τη φύση της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις, στη δεύτερη ερώτησή σας για την προστασία από κερδοσκόπους. Εδώ δεν θέλω να κάνω και άλλα σχόλια πέρα αυτών που έχω ήδη κάνει. Έχω πει ότι είναι ένα γενικό ζήτημα αυτό το να διασφαλίζουμε την ε, σωστή λειτουργία των αγορών και σε αυτό θα μείνω. Στην ειδική περίπτωση, κάθε φορά που υπάρχει ειδική περίπτωση πρέπει να εξετάσουμε την ειδική περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο ότι αν έχουμε μια ισχυρή θέση και σαφή θέση, πιστεύω ότι οι εντάσεις θα διαλυθούν. Χρειάζεται βέβαια πειθαρχία, πειθαρχία προς όλους. Και στην Ελλάδα. Και για το τελευταίο, για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που χρειαζόταν από την αρχή ήταν η εμπλοκή των ίδιων των κυβερνήσεων. Τα μέσα τα έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ δεν νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρώνεται στην αλλαγή των θεσμών, των οργάνων, να φτιάχνει καινούργιες ρυθμίσεις κλπ. Όχι, αυτό που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα από τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι που διακυδεύεται εδώ. Να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνη οι κυβερνήσεις. Και η παρούσα εμπειρία μας βοηθάει σε αυτό, γιατί μας αναγκάζει όλους να φροντίσουμε να αναλάβουμε στο επακρό τη ευθύνε μας. Ευχαριστώ, ο κύριος Γκαρθία Μαργάγιο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για την εποπτεία στο ελληνικό, στο έλλειμμα, στις ε, παγκόσμιες ανισορροπίες, όπου βλέπουμε να παίζεται εδώ το έλλειμμα του κινέζικου νομίσματος. Βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα, τι θα κάνει. Τι θα κάνει η τράπεζα άμα οι Κινέζοι αρχίζουν να ξεφορτώνονται τα αποθέματα τους σε δολάρια. Επίσης, ξέρουμε ότι λειτουργήσε άσχημα το θέμα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι αυτά τα 14 σχέδια σταθερότητας ήταν καθαρά γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε άλλα κριτήρια, ας πούμε να έχουμε έλλειμμα ανατρέχοντα λογαριασμό ή άλλα κριτήρια για να μπορούμε να βγάλουμε ακριβώς το τι γίνεται στα κράτη-μέλη. για το 2004, για το 2005 ξέραμε ότι δεν θα εφαρμοζόταν ποτέ το σύμφωνο σταθερότητας κυρίως για τους μεγάλους, δεν ξέρουμε και για τους μικρούς τι θα γίνει. Λοιπόν, μήπως θα έπρεπε εμείς να αφήσουμε τις κυρώσεις έτσι όπως έχουμε και να, περιορίσουμε την πρόσβαση στα μερίδια του προϋπολογισμού υπολογισμού ως ποινή. Εσείς επίσης πιστεύετε ότι, τρίτη ερώτηση, ότι αυτή η λεγόμενη κερδοσκοπική δράση των τραπεζών έναντι της Ελλάδος και η χειραγώγηση που έκανε η Ελλάδα στους λογαριασμούς της, η λεγόμενη χειραγώγηση. Τι λέτε εσείς, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έγινε, χρειαζόταν περισσότερη εποπτεία, πώς θα λειτουργούσε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο για τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Αυτές ευθύνονται για την τραγική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε διεθνώς. Εάν δεν υπάρξει αποτελεσματικότητα στην εποπτεία που γίνεται σε επίπεδο της ομάδας των 20, του G20, οι οικονομίες, κυρίως εκείνες που σε διεθνές επίπεδο έχουν ανισορροπίες, θα μας οδηγήσουν σε νέα κρίση. Άρα δεν φτάνει να πάρουμε μαθήματα από τις δημοσιονομικές αγορές, αλλά και από τις μακροοικονομικές πολιτικές των ε, χωρών που ευθύνονται για τις μεγάλες ανισορροπίες, είτε πρόκειται για πλεονάσματα, είτε πρόκειται για λύματα. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η θέση της Ευρώπης σε σχέση με την Κίνα την τελευταία συνάντηση των 20 επαναλάβαμε αυτό που είπαμε και στην Κωνσταντινούπολη. Ότι δηλαδή χρειάζεται μια ε, προδευτική αντιμετώπιση του νομίσματος της Κίνας που θα συνεισφέρει στην ισορροπία διεθνώς. Όσον αφορά τώρα το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, για άλλη μια φορά κάνω έκκληση για την εφαρμογή του. Έχει αποφασιστεί το σύμφωνο, έχει αναθεωρηθεί, έχει πια μπει για τα καλά στη συνθήκη και ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει αν δεν το εφαρμόζουμε. Δεν ζητάω αλλαγή του, αλλά ζητάω εφαρμογή του. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να το εφαρμόζουμε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια πολύ ισχυρή έκκληση προς την κατεύθυνση αυτή, να το εφαρμόσουμε. Και δεν θα έλεγα ξεχάστε τις κυρώσεις, όχι. Είναι αλήθεια ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Είναι αλήθεια επίσης ότι αντισταθήκαμε, ότι είπαμε ότι δεν θα έπρεπε. Θυμόσαστε, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τσακωνόντουσαν. Πήγανε στο δικαστήριο. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο σήμερα παραποτέ η ιδέα αυτή ότι το σύμφωνο πρέπει να εφαρμόζεται και να επιβάλλονται και κυρώσεις σε αντίθετη περίπτωση είναι το σωστό. Βέβαια, είμαστε σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που φαίνεται να είναι αδύνατο κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι λέω ότι εμείς αυτό ζητάμε. Και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να κάνουμε. Μην είμαστε κοντόφθαλμοι σήμερα. Για το τελευταίο. Η Eurostat πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει επιτόπου και να μπορεί από κοντά να πάρει ό,τι πληροφορίες χρειάζονται και να είναι σίγουρο ότι υπάρχουν οι πληροφορίες που χρειάζονται και να επιμείνει για αυτές. Δεν μπορούμε να δεχτούμε στο μέλλον να έχουμε τέτοιες ε, παρατυπίες ουσιαστικά που οδηγούν σε μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας. Κάτι τέτοιο έχει τραγικές συνέπειες και καταστρέφει την αξιοπιστία. Επιμένω σε αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να το γνωρίζουν. Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν ε, μερικές φορές ε, δεν ήμασταν πρόθυμοι για ομές αποφάσεις. Τώρα πρέπει να το κάνουμε. Παρακαλώ. Η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Διοικητά, υπάρχουν δύο ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένες. Πρώτο ερώτημα. Θεωρείτε ότι χρειάζεται ένας αυστηρά ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης μιας χώρας η οποία αντιμετωπίζει ακραίες οικονομικές δυσχέρειες όπως η αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, θεωρείτε ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός υπό ποιες συνθήκες. Και επίσης το ποσοστό 6,25 ως επιτόκιο που προσφερόταν στην Ελλάδα για το δανεισμό της στις αρχές Μαρτίου που ήταν τόσο ακραίο δεν μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Δεν θα ε, δικαιολογούσε δηλαδή την ε, θέση σε λειτουργία ενός τέτοιου μηχανισμού. Ευχαριστώ. Κύριο Τρισέ, ευχαριστώ. Δεν θα επανέλθω στα όσα είπα νωρίτερα. Ανέφερα νωρίτερα τους όρους που θεωρώ απαραίτητους για την προσφορά ενός τέτοιου συνόλου συνθήκων. Όπως νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον τους όρους του Συμβουλίου, δηλαδή χωρίς ειδικέ ε, δεσμεύσεις, ε, χωρίς επιδότηση δηλαδή, στήριξη από πλευράς του Συμβουλίου. Είπαμε ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι πολύ αυστηροί, δεν θα υπάρχει χαρακτήρας δωρεάς, θα είναι άκρος ε, κατεπίγουσα η κατάσταση και θα υπάρχει άμεσος κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος για το ίδιο το κράτος μέλος και για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. Και οι τρεις όροι πρέπει να υπάρχουν. Ο κύριος Σκούτας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δίκητα. Μιλούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις έννοιες της αλληλεγγύης, της ευθύνης, της επιτήρησης. Μέτρα τα οποία εγώ θα χαρακτήριζα ήπια μέτρα. Υπάρχουν λοιπόν τίποτα πιο σκληρά, όχι το software αλλά το hardware, το υλικό θα λέγαμε. Τίποτε πιο απτό, φερρυπίν, κάποια ε, πιο συγκεκριμένη δομή της φορολογικής διακυβέρνησης στο μέλλον που να καλύπτει όλους τους παράγοντες και τις κεντρικές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στους κόλπους της. Αυτό το αρχιτεκτόνημα για το μέλλον πώς το βλέπετε εσείς να διαμορφώνετε. Τρισέ. Πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι οι οργανισμοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο καθένας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως καθήκον την αξιοπιστία στην εξασφάλιση σταθερότητας των τιμών πρόθεσμα, στην ε, ικανοποίηση των προσδοκιών δηλαδή με τη σταθερότητα των τιμών να, υπάρχει αυτή η προσδοκία, η, βεβαιότητα για τον Ευρωπαίο μιας ε, βιώσιμης ανάπτυξης, διατήρησης εργασίας του, οικονομική σταθερότητα, νομισματικής ε, σταθερότητας. Ευθύνη τη κυβέρνηση του, από την άλλη, είναι να εξασφαλίσει την φορολογική πολιτική που θα εμπνέει εμπιστοσύνη, που δεν θα επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές, τα παιδιά και τα εγγόνια, που δεν θα θεωρηθεί αναξιόπιστη από τους πάντες, πολίτες δηλαδή και οικονομικούς φορείς, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η οικονομία και η θέση εργασίας. Και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη αλλά και στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα υπάρχει η επιτήρηση των αδελφών κυβερνήσεων που έχουν επίσης τη δική τους ευθύνη, όπως το αποφάσισαν οι λαοί της Ευρώπης. Γιατί οι λαοί της Ευρώπης ήταν αυτοί οι οποίοι απεφάσισαν αυτή τη λειτουργία της επιτήρησης δυνάμει των συνθήκων και, σταθερό, και του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Υπάρχει το hardware στο οποίο αναφερθήκατε, το υλικό δηλαδή τα τα μέτρα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε να πούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη χειρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ίσως χειρότερη ακόμη εν δυνάμει από αυτήν που ακολούθησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πράγμα βέβαια το οποίο δεν βοηθάει καθόλου κανέναν από του οργανισμού που έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα, ούτε τι εθνικέ κυβερνήσει, ούτε τα κοινοβούλια, ούτε και του ε, εκπροσώπου που βρίσκονται μέσα στο Συμβούλιο, δηλαδή του ομολόγου, το Συμβούλιο ω συλλογικό όργανο. Δεν υποτιμώ το έργο που έχει αναλάβει ο καθένα από αυτού του φορεί αλλά παρακαλώ μην υποτιμούμε το εφιστάμενο hardware. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει το hardware, αρκεί για να κάνει τη δουλειά του. Κύριε Σμέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, μιλήσατε για τον κοινό προορισμό, όχι μόνο των χωρών μέσα στην Ευρωζώνη όμως, έχει να κάνει με ολόκληρη την Ευρώπη και με τις 27 χώρες μέλη. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη και πολύ θα ήθελα να μπαίναμε και εμείς στην Ευρωζώνη. Το 2008, το 2009 μπορούσε κανείς αυτό να το εξηγήσει εύκολα και σε όποιον το έλεγα ε, δεν είχε επιχειρήματα να αντιπαραθέσει. Τώρα όμως έχουν αντεπιχειρήματα, μου υπενθυμίζουν και το δημοψήφισμα που είχαμε το 2003 και λένε ότι δεν είναι η καλύτερη νομισματική ζώνη. Μου λένε δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Θα λειτουργούσε μόνο αν υπήρχε και φορολογική ένωση. Εσείς τι επιχειρήματα υπέρ της Ευρωζώνης μπορείτε να μου δώσετε σήμερα κύριε Τρισέ, για να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω κι εγώ. Η Ελλάδα Χωρίς το ευρώ αν είχε μείνει απ' έξω, τι θα είχε χάσει η Ευρωζώνη. Σήμερα λοιπόν, για να είναι κανείς μέλος της Ευρωζώνης, τι έχει να κερδίσει. Μπορείτε να μου πείτε. Τρίσε, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολη η ερώτηση. Όταν δημιουργήθηκε η ιδέα, ήταν ξεκάθαρο ότι επιπλέον από την εποπτεία που θα γινόταν μέσα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με ακούσατε πριν που, είπε, που είπα και επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση πρέπει να είναι και νομισματική και οικονομική δεν μπορεί να είναι μόνο νομισματική, πρέπει να είναι και οικονομική. Και στην καρδιά της οικονομικής βρίσκεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Από την αρχή λοιπόν που σχεδιάστηκε η ιδέα αυτή, το βασικό ήταν ότι θα βοηθούσε η πίεση μεταξύ ομοτήμων. Η πίεση από την ίδια την ευρωζώνη του ενός πάνω στον άλλον. Συνεπώς, ότι θα ήταν καλό να μην συγχωνευτούν όλα τα δημοσιονομικά. Αυτό το αποφάσισαν οι ίδιοι, οι ιδρυτές. Και αν ε, θέλω να είμαι θετικό, θα πω ότι η Ελλάδα ήταν σε πολύ ε, κακή κατάσταση. Η πίεση όμως των ομοτήμων, ιδιαίτερα στο τελευταίο συμβούλιο, συν η πίεση της αγοράς, οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση που εγώ ο ίδιος ονομάζω πιστική και θαραλέα. Δηλαδή αυτό που έχετε μπροστά σας σήμερα είναι ένα επεισόδιο στην λειτουργία αυτού που από την αρχή οι ιδρυτές θεώρησαν μηχανισμό με δύο σκέλη. Μηχανισμό, μηχανισμό πίεσης με δύο σκέλη. Σήμερα βλέπουμε ότι ένα μέρος της αγοράς είναι διστακτικό. Για μένα είναι μεταβατικό αυτό, διότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση, που είναι θαραλέες και πιστικές, είναι τέτοιες που θα αναγνωριστούν τελικά. Από εδώ και πέρα βέβαια θα δούμε τι θα συμβεί. Και επιπλέον υπάρχει και η αίσθηση που έχει εκφραστεί από τους επικεφαλείς και θα σας το ξαναδιαβάσω γιατί υπάρχει, το υπέγραψαν οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει συντονισμένη δράση εφόσον χρειαστεί γιατί υπάρχει απειλή για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή εδώ έχετε την σωστή αντίδραση και τη σωστή απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Επιπλέον μπορείτε να πείτε ότι η παγιωμένη θέση της Ευρωζώνης είναι καλύτερη από ε, άλλες περιπτώσεις, από τους 7 για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι που δείχνει πολύ δυνατό. Η κατάσταση για την ελληνική κυβέρνηση μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, αλλά συγχρόνως υπάρχει σχεδιασμός για τη λειτουργία της Ευρωζώνης, ακόμα και σε στιγμές δύσκολες. Όμως εγώ είμαι αισιόδοξο. Γκέι Μίτσελ και παρακαλώ να μην ξεχνάτε ότι έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε πέντε λεπτά καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, πριν από δύο χρόνια νομίζω σας είχα ε, θέσει το ζήτημα των υπερβολικών πληθωριστικών πιέσεων σε σχέση και με τις ε, φούσκες στην αγορά. Ίσως λοιπόν τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε κάτι άλλο. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα του συμπολίτε μου, του ψηφοφόρου στη δική μου εκλογική περιφέρεια, ιδιαίτερα αλλά και τη χώρα μου γενικότερα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν σε αυτόματο πιλότο, νομίζω, και γι' αυτό έχουμε αντιμετωπίσει όλε αυτέ τι δυσκολίε. σω ήταν διαφορετικά τα πράγματα εάν δεν είχαμε αυτόματο πιλότο. Εάν λοιπόν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει μπορούσαν να δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία, μία ή δύο η κάθε μία στην Ευρώπη ολόκληρη, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Έτσι πιστεύω. Το πρόβλημα όμω είναι ότι έχουμε, ε, έχουμε ως διαχειριστεί μια τράπεζα. Η Την τράπεζα ως ιδέα δηλαδή. Η τράπεζα έχει μάθει τον κίνδυνό τη να τον υπολογίζει με βάση το κέρδος το οποίο μπορεί να προσμένει να εξασφαλίσει. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κάνει τον υπολογισμό του αν θα δώσει δάνειο και τι είδους, τι είδους, τι είδους κίνδυνο αναλαμβάνει με βάση τον άνθρωπο στον οποίο θα χορηγήσει το δάνειο. Πρέπει να τον γνωρίζει αν θα είναι ικανός, αν θα κάνει καλά τη δουλειά του, αν θα μπορέσει να την ξεπληρώσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και θέλω εδώ, γιατί δεν θέλω να φύγω και να κάνω μια ερώτηση μόνο για τον πληθωρισμό και να πούμε ότι έληξε το θέμα, για το σύστημα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ίδια. Δεν θα έπρεπε να γυρίσουμε στην παλιά ιδέα του τραπεζίτη, ο οποίο ξέρει να κάνει τη δουλειά του, που γνωρίζει τον πελάτη του και που υπολογίζει τον κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνει με το δάνειο που θα δώσει. Τρισε, θα συμφωνήσω πολύ μαζί σα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η σοφία, η εμπειρία του κλασικού εμπορικού τραπεζίτη, αυτή τη δομή που σήμαινε ότι μπορεί κανεί να υπολογίσει τον κίνδυνο και ιδιαίτερα για τη μεσαία και τη μικρή επιχείρηση. Είναι καθοριστική σημασία και είναι και ο λόγο για τον οποίο οι ελεύθερε οικογενειακέ αγορά έχουν αυτή την την ε, διάσταση της τράπεζας δηλαδή και έχουν θέσει την τράπεζα να υπολογίζει τον κίνδυνο και τις επιτρέπουν τις κάθε τράπεζας να, να επιλέγει και να μην είναι υποχρεωμένα να λέει ναι την εποχή των παγιών αγελάδων και όχι την εποχή των ισνών αγελάδων, είναι ακριβώς αυτή η ιδέα ότι προσαρμόζεται η τράπεζα στην, ε, στις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς και στον πελάτη που θα έχει. Δεν υπάρχει ε, μία συνταγή για τους πάντες, όπως δεν υπάρχει καμία τράπεζα που να καλύπτει όλες τις ανάγκες όλων των πελατών και δεν υπάρχει και ενία εικόνα του πελάτη. Ασφαλώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο χρηματοπιστωτικό μα σύστημα, στο τραπεζικό μα σύστημα, σε όλη τη ζώνη του ευρώ, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ πολύ μαζί σα. Η κυρία Λούλινγκ, από ό,τι φαίνεται, εξαφανίστηκε προσωρινώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Γκέμπερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εσείς επιμείνατε πολλές φορές στην, ε, στους όρους για τη χορήγηση δανείου στα κράτη-μέλη. Από την κρίση και μετά η Κεντρική Τράπεζα έπαιξε πολύ σωστά το ρόλο της δανειοδοτώντας και με, ε, και ένα επιτόκιο ιδιαίτερα ευνοϊκό. Όπως είπατε μια άλλη φορά δεν ζητήσατε καν την ταυτότητα των τραπεζών που ερχόντουσαν να χρηματοδοτούν. Αλλά όμως εσείς αναρωτηθήκατε αν τα χρήματα που πήραν οι τράπεζε από εσά δεν τα χρησιμοποίησαν για να κερδοσκοπήσουν στο νομισματικό, στην, νομισματική αγορά. Εσεί είστε ένα θεσμικό όργανο, έχετε την Ευρωμάδα απέναντί σα από εσά, η οποία όμως είναι μια συσπήρωση κρατών μελών, μια συνένωση κρατών μελών, χωρίς ε, εσωτερική αλληλεγγύη μέσα στην Ένωση επίσης, πολύ χαμηλότερος προϋπολογισμός από ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός των κρατών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε πέντε διαφορετικές χρηματιστηριακές αγορές τουλάχιστον. Εσείς φανταστήκατε να δημιουργήσετε ποτέ μία κοινή αγορά ευρωομολόγων που θα βοηθούσαν πολύ περισσότερο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για το πρώτο σημείο πρέπει να σας πω ότι έχουμε κανόνες ε, για την χρηματοδότηση των τραπεζών. Πρέπει αυτές οι τράπεζες να πληρούν αυτούς τους κανόνες. Εμείς δεν κάνουμε άλλον έλεγχο πέρα από αυτόν που ασκούν όλοι οι οργανισμοί ε, τραπεζικής εποπτείας, είτε είναι τράπεζες του ευρωσυστήματος, είτε είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί εξαρτάται τις χώρες. Λοιπόν, αυτή, αυτή λοιπόν η εποπτεία ασκείται από τους υπεύθυνου. Λοιπόν, εμείς πρέπει απλώς να έχουμε εγγύηση για τη ρευστότητα των τραπεζών. Εγώ είπα στην εισαγωγή μου ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις ε, αρχίζουν και περιορίζονται για να περάσουμε σε μια κατάσταση πιο νορμάλ. Για τη δεύτερη παρατήρηση όντως αληθεύει η Ευρωζώνη οικοδομήθηκε αφήνοντας ε, τα κράτη ε, να είναι υπεύθυνα για τη δική τους δημοσιονομική διαχείριση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς είπαμε πάντοτε αυστηρή παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για το ενιαίο νόμισμα και επίσης εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών και των εξελίξεων του κόστου σχετικής ανταγωνιστικότητας που συνδέονται. Διότι αν αφήσετε να καλπάζουν οι μισθοί και οι αμοιβέ ε, στο δημόσιο τομέα, τότε εσείς μειώνετε το σχετικό σας ανταγωνισμό και διαλύετε την οικονομία σας. Αλλά δεν θα εκπλαγείτε άμα σας πω ότι δεν είμαστε υπέρ εκδόσεων ευρωμολόγων, κοινών ευρωμολόγων, διότι τότε εδώ μπερδεύουμε όλες τις δημοσιονομικές πολιτικές, σίγουρα μπορεί να υπάρξουν όσον αφορά στη ρευστότητα, να υπάρξουν πλεονεκτήματα. Αλλά θα υπάρξει ένα μεγάλο μειονέκτημα, δεν θα γίνεται πλέον διαφορά μεταξύ μιας καλής διαχείρισης και μιας κακής διαχείρισης. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ένα ολοκληρωμένο ομοσπονδιακό σύστημα, δεν είναι απαραίτητα σωστό να μην κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ της εύνομης διαχείρισης και της μη εύνομης διαχείρισης. Έτσι λοιπόν εμείς δεν είμαστε υπέρ ε, της έκδοσης ευρωτήτλων με μια κοινή υπογραφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στις παγκόσμιες ανισορροπίες και είπατε ότι έχουν μεγάλη σημασία για τη σημερινή κατάσταση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για τις μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τις ανισορροπίες αυτές. Ένας από τους κύριους παράγοντες για την σημερινή δημοσιονομική κρίση ήταν ακριβώς η συσσόρευση ανισορροπιών στην αγορά κινήτων. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα περιοριστώ στις ερωτήσεις μου, θα τις κάνω εύκολες. Πρώτον, οι κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσαν να δουν τις εξελίξεις των τιμών στα κίνητα περισσότερο να τις λάβουν υπόψη τους δηλαδή για τις μελλοντικέ τους πολιτικές. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακούσει τη φωνή διάφορων εμπειρογνωμόνων και θα λάβει υπόψη τις, τις θέσεις τους όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων για να προσαρμόσει τους δείκτες τιμών. Και τρίτον, θα ληφθούν υπόψη οι ανισορροπίες αυτές περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας που είναι πολύ σημαντικές. Πρώτον, θα έλεγα ότι έχετε δίκιο για το ότι τα κίνητα και η φούσκα των ακινήτων έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα διάφορα μπούμ που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε. Και πόσο ξέρω, όλες οι τράπεζες ε, ψάχνουν να βρουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι τα κίνητα είναι υπεύθυνα κυρίως για τις φούσκες αυτές. Και η συζήτηση δεν είναι καταδημαϊκή. Όλες οι τράπεζες στον κόσμο ασχολούνται με αυτό, αλλά βέβαια οι υπεύθυνοι δεν καταλήγουν εύκολα σε μια απάντηση. Οι συμπεριφορές είναι διαφορετικές η εμπειρία που έχει κανείς ε, διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Οπότε δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι θα σταθεροποιήσουμε τις ε, τιμές των κατοικιών αυτόματα. Και στην Ευρώπη βλέπετε ότι γίνονται προσπάθειες, αλλού είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το CPI. Πώς θα περιορίσουμε δηλαδή τις φούσκες αυτές με διάφορα μέσα. Εξακολουθούμε να το συζητάμε, να προσπαθούμε να βρούμε λύση. Έχει γίνει συζήτηση στην Κεντρική Τράπεζα και με την Eurostat. Υπάρχουν διάφορες σχολές από αυτού. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών, ο σημερινός που έχουμε, είναι κατά πάσα πιθανότητα ο καλύτερος δείκτης που μπορούμε να προσφέρουμε. Αλλά δέχομαι ότι ναι μεν είναι το καλύτερο που έχουμε να προσφέρουμε, αλλά θεωρητικά δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να υπάρχει. Όπως βλέπετε είμαι πολύ προσεκτικός στην απάντησή μου. Είχατε και κάτι τρίτο Απάντησα στην τρίτη σας ερώτηση, ρωτά ο κύριος Τρισέ. Να λάβετε υπόψη σας τις ανισορροπίες αυτές στο μέλλον. Θα τις λάβετε υπόψη σας και πώς. Απάντησε ο κύριος Τρισέ. Ναι, ναι, βέβαια. Όπως ξέρετε, το γεγονός ότι εξετάζουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε από τα νομισματικά δεδομένα, όλους τους παράγοντες, έχετε έτσι τις πιστώσεις για τα κίνητα. Τις εξετάζουμε και αυτές πάρα πολύ προσεκτικά. Το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις τύπου, πολλές φορές και στο Κοινοβούλιο, ότι η ένδειξη που έχουμε συνάδει με αυτά που αντιλαμβανόμαστε και εμείς όταν παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τα επιτόκια. Τις λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν. Ε, μας βοηθήσουν οι διερμηνείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε άλλα 10-15 λεπτά. Κυρία Λούλινγκ, γυρίσατε βλέπω, είχατε χάσει το, τη σειρά σας, αλλά ξανά ήρθατε. Ε, ναι, μα πρόεδρε, είχα καταλάβει ότι δεν είχα το δικαίωμα να υποβάλω ερώτηση στον κύριο Τρισέ γι' αυτό. Ε, έχω την εξή ερώτηση λοιπόν, διότι ο πρόεδρος της Eurogroup αναφερόμενος στην ε, ιδέα του μηχανισμού για προσφορά βοήθεια στην Ελλάδα, είπε ότι ασφαλώς δεν υπάρχουν διμερείς εγγύησεις, όμως μίλησε για διμερή βοήθεια. Μπορείτε λοιπόν κύριε Τρισέ να μου εξηγήσετε γιατί ορισμένες χώρες δεν συμμετέχουν στις διμερείς εγγυήσεις προς την Ελλάδα και αυτές οι ίδιες χώρες μήπως δεν, συμμετέχουν, δεν συμμετάσχουν ούτε στη διμερή βοήθεια. Γιατί δεν βλέπω ακριβώς που έγινε η διαφορά μεταξύ διμερών εγγυήσεων και διμερούς βοήθειας. Εάν κάποιος δεν θέλει να προσφέρει διμερή εγγύηση, πώς μπορεί να θέλει να προσφέρει διμερή βοήθεια. Πώς το βλέπετε σε αυτό. Τρισέ. Καταρχάς, εγώ δεν θα την χαρακτηρίσω αναγκαστικά ως βοήθεια, γιατί όπως έλεγα δεν χρειάζεται να υπάρχει στοιχείο επιδότησης στα όσα γίνονται. Όχι λοιπόν ειδική μορφή δάνεια, όχι επιδότηση. Ο πρόεδρος της Eurogroup μιλάει για τα θέματα της δικής του ευθύνης και αρμοδιότητας, δηλαδή την αναρμόνιση των αποφάσεων που λαμβάνουν διάφορες χώρες. Εγώ πάλι δεν έχω αυτή την αρμοδιότητα, αν μου επιτρέπετε να το σημειώσω. μόνο μπορώ να σας πω είναι οι όροι τους οποίους θεωρώ εγώ απαραίτητους για την ανάπτυξη των συνθήκων ε, που θα χρειαστεί να υπολογιστούν. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω κάποια στοιχεία μη ε, μορφής, όχι επιδόσεις δηλαδή, στα οποία θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, όπως αυτό αναφέρεται στο ανακοινωθέν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Αλλά ο κύριος πρόεδρος της Eurogroup, ο Jean-Claude Juncker, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσει αυτήν την ερώτηση, γιατί δική του αρμοδιότητα είναι. Η πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. ήταν ο πρώτος και ο μόνος ε, που είχε την ευκαιρία. Ε, κύριε Τρισέ, πολύ σύντομα για τις ανισορροπίες. Είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα προ ανισορροπίε αλλά και για ορισμένε χώρε που έχουν πλεόνασμα, πλην όμω όχι για τη Γερμανία που έχει μεγάλο δημογραφικό ζήτημα. Όμω, αν κοιτάξουμε του ε, τρέχοντες λογαριασμούς καταλήγουμε στο συμπεράσμα, όπως είπατε, ότι θα πρέπει να αποταμιεύουμε περισσότερο. Όμως δημογραφικό πρόβλημα, οι δυσκολίες δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει να αφήσουμε το κόστος του εργατικού δυναμικού να αναπτυχθεί σε επίπεδα κάτω από τους στόχους Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά δεν καταλαβαίνω την εξήγηση που δώσατε. Και παρακαλώ να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις για όσους θεωρούν ότι θα πρέπει η Ευρώπη να συμπεριφέρεται κατά τρόπο πιο φιλοευρωπαϊκό. Από ό,τι τουλάχιστον φάνηκε να λέτε εσείς δημοσίως. Και από ό,τι φαίνηκε να έχετε κάνει και ακόμη πιο σκληρούς όρους σε, στο εσωτερικό των συνεδριάσεων, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών. Απάντηση, για να συνοψίζουμε. Εάν κρίνει κανείς το επίπεδο των ε, ισοζυγίων, τρεχόντων λογαριασμών ή των πλεονασμάτων θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη τι δημογραφικές συνθήκες μιας χώρας, χώρας και είναι τεράστιες οι διαφορές ό,τι και να πούμε. Άρα δεν λέω ότι μπορεί όλο το πλεόνασμα της Γερμανίας να εξηγηθεί από τις δημογραφικές πιέσεις, αλλά μεγάλο μέρος του ναι και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Δεύτερον, και όσον αφορά το κόστος της ανταγωνιστικότητας, ε, το κόστος μάλλον της, ε, του εργατικού δυναμικού, ναι όντως, η Γερμανία ξεκίνησε με ανταγωνιστικό, ανταγωνιστική σχέση δυσμενή. Είχε λιγότερο δηλαδή ε, καλή θέση στην αρχή τουλάχιστον της ένταξης στο ευρώ, αρχή της εισαγωγής στο ευρώ, λόγω των συνθήκων της επανένωσης. Όπως είπαμε ήταν λιγότερο ανταγωνιστική η θέση της. Τώρα, όπως λέτε, θα μπορούσα λίγο πολύ να συμφωνήσω ίσως ότι αυτή η ανταγωνιστικότητα μέσα στην ζώνη του ευρώ έχει καλύψει πλέον η Γερμανία την ανταγωνιστικότητα της, άρα δεν χρειάζεται να καλύψει άλλο έδαφος στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον και θα πρέπει πλέον να λάβουμε υπόψη το δικό μας το όριο που έχουμε ορίσει, τον προϋπολογισμό, δηλαδή το 2 το πολύ μέσα στη ζώνη του ευρώ, σε 100 βέβαια, μεσοπρόθεσμα, γιατί μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψει, αλλά θα μπορούσαμε μεσοπρόθεσμα να δούμε μια διακύμανση για τις οικονομίες αυτές και όχι μόνο τη Γερμανία, οι οποίε θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι η σχετική του ανταγωνιστικότητα μέσα στη ζώνη του ευρώ είναι λίγο πολύ ικανοποιητική. Όχι, εν πάση περιπτώσει, τελείω με, με μεγάλες ανισορροπίες. Αυτό για τις χώρες που έχουν μια κάποια ε, ισορροπία στην ανταγωνιστικότητά τους. Έτσι μπορούμε να αναλύσουμε με βάση τα, τα δημογραφικά στοιχεία, την σχετική ανταγωνιστικότητα, την ε, εξασφάλιση μεριδίου αγοράς ή την απώλεια μεριδίου αγοράς μέσα στη ζώνη του ευρώ και βεβαίως και άλλες πιθανές έννοιες και κριτήρια. Αλλά βλέπετε τι εννοώ εγώ με, την, με τις κρίσεις τις οποίες διατυπώνω, διότι αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι μόνο να μιλήσω εκ μέρου των 16 ε, των 16 κρατών των 330 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης που είναι στη ζώνη του ευρώ. Η πρόεδρος, ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται τα λεφτά μας πιάσαν τόπο ή μάλλον το έλλειμμά μας έπιασε τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπατε. Με συγχωρείτε αν ήμουν πότε αυστηρή και πότε ε, λιγότερο αυστηρή ως προς την τήρηση του χρόνου. Ευχαριστούμε τους Ερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Οι Ερμηνείς σας ευχαριστούν. Μερικές φορές, ε, για να μην σας καθυστερώ τώρα, ε, θα σας πω ότι αύριο το πρωί ξεκινάμε 9.30 το πρωί, γιατί βλέπω ότι όλοι φεύγουν.